I think we can start. Μπορούμε να ξεκινήσουμε. Το χειρότερο. Κράμερ εδαγίων κράμερ. Αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίε και κύριοι, ξεκινάμε τη συνεδρίασή μας. Η μερίσια διάταξη γίνεται δεκτή εκτό αν έχετε κάποια αντίρρηση. Όχι. Δεν έχω καμία ανακοίνωση ως πρόεδρος. <clears throat> Μπορούμε να περάσουμε κατευθείαν στο σημείο 3. Task Force για τον τουρισμό και Ευρωπαϊκή Τουριστική Πολιτική. Έχουμε ανταλλαγή απόψε με τον κύριο Πέτρο Ορτούν από τη Γενική Διεύθυνση έντρα. Ερχόμαστε λοιπόν στην πρώτη συνεδρίαση της ε, Task Force μετά από την ε, ε νέα θητεία μας, της Κομισιόν. Ο κύριος ε, ο Ουιχέη είναι ο αντιπρόεδρος της ε, Task Force, της Ειδική μονάδας για τον τουρισμό και χαιρόμαστε για την παρουσία του και ο κύριος Πέδρο Ορτούν έχει προσκληθεί να μας δώσει μια γενική επισκόψη για την κατάσταση της ευρωπαϊκής πολιτικής τουρισμού. Με μεγάλη χαρά σας καλωσορίζω κύριε Ορτούν και χαίρομαι πάρα πολύ για το γεγονός ότι συμπίπτει η παρουσία σας με την ε, ανακοίνωση της νέας πρωτοβουλίας της Κομισιόν και μάθαμε ότι η Επίτροπος Μπιενκόφσκι έχει αναφέρει μια σειρά από κοινέ δράσεις οι οποίες θα είναι και αντικείμενο μια ανακοίνωσης της Κομισιόν το, φθιν, το φθινόπωρο. Με τον τρόπο αυτό θα δημιουργηθεί ένα νέο πλαίσιο για τον ευρωπαϊκό τουρισμό και θα υπάρξει ένα πακέτο 10 δράσεων που ήδη έχει δημοσιευτεί από το 2010. Ο τίτλος του είναι φιλόδοξος «Η Ευρώπη ο καλύτερος τουριστικός προορισμός του κόσμου» και φυσικά θα αποτελέσει αντικείμενο μιας έκθεσης που θα εκπονήσει η κυρία Φιντάντσα. Ε, χαίρο, χαίρομαι λοιπόν για την παρουσία σας και θα ήθελα να μας δώσετε πληροφορίες όχι μονάχα για το νέο αυτό πακέτο, αλλά <clears throat> και να μας αναφέρετε για τη συνέχεια που έχει δοθεί στις δράσεις οι οποίες ξεκίνησαν το 2010. Έχετε το λόγο κύριε Ορτούν. Ευχαριστώ. Καλημέρα σας όλοι. Ναι, όπως είπατε και θα σας ενημερώσω γύρω από δύο άξονες σε σχέση με το τι κάναμε μετά την ανακοίνωση του 10. Έχουμε τώρα την κυρία Βινκόφσκα που είναι η νέα μας επίτροπος και πριν από δύο ε, μέρες στη Μαδρίτη τρίτη πρωί ανακοίνωσε και υποσχέθηκε που ίσως το ξέρετε το, ίσως παρακολουθήκατε από το ίντερνετ κατόπιν των ακροάσεων της Δευτέρας Οκτωβρίου είπε έλεγα ότι κατόπιν μια σειρά διαβουλεύσεων όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς ιδιωτικοί και δημόσια πρόκειται να συμμετάσχουν σε κάποιες κοινέ δράσεις τόσο ώστε να είναι ο ευρωπαϊκός τουρισμός πιο ανταγωνιστικός και να έχουμε κάποιο είδους αηφόρα βιώσιμη ανάπτυξη στην δραστηριότητα αυτού του κλάδου. Έτσι έχουν τα πράγματα. Επομένως νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό και τέλος πάντων μεγάλη μου χαρά να έρχομαι εδώ να συζητώ μαζί σας για αυτά τα ζητήματα που αφορούν την πολιτική του τουρισμού. Από ό,τι ξέρω έχουμε μια φρέσκια φουρνιά από ευρωβουλευτές και θα πρέπει σε εκείνους ιδίως να υπενθυμίσω ότι από το 2009 συγκεκριμένε αρμοδιότητε δύναμη τη Λισαβόνα. Πρόκειται για αρμοδιότητε τρίτου επίπεδου. Οπότε η Ευρωπαϊκή Ένωση πρόκειται και δύναται να υποστηρίξει με κάθε είδου μέτρα τις προσπάθειες για να υποστηρίξει δηλαδή τις προσπάθειες των κρατών μελών. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό και άρα πρέπει να εναρμονίσουμε την νομοθεσία τη σχετιζόμενη με τον τουρισμό. Άρα θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να προσδώσει αυτού του είδους την προσθεμένη αξία σε αυτή την νομοθεσία και έτσι να έχει ο τουρισμός μας. Θα θυμάστε ότι όταν έλαβε το Φεβρουάριο του 2010 ο σημερινός σας αντιπρόεδρος κ. Σταγιάννη είχε δημοσιεύσει αυτήν την ανακοίνωση και τον Ιούνιο εγκρίναμε 21 δράσεις οριζόντιες ούτως ώστε ο τουρισμός να γίνει αντικείμενο mainstream δηλαδή να ενταχθεί σε όλες τις άλλες ευρωπαϊκές πολιτικές. Αλλά και σε όλα τα χρηματοοικονομικά μέσα πολιτικής της Ένωσης. Τελευταία τέσσερα χρόνια ακριβώς αυτό κάναμε και εμείς. Αυτές τις 21 δράσεις τις προχωρήσαμε. Έτσι θέλουμε τα προϊόντα τουρισμού να είναι πολύ μορφή στην Ευρωπαϊκή Ένωση και είπαμε ότι να έχουμε προπαρασκευαστικές δράσεις, πιλωτικά προγράμματα, τα γνωρίζετε κύριε Κράμερ. όπω το ICT, πολιτιστικά προϊόντα, προϊόντα τουρισμού. Είχαμε τη δράση Καλυψό το 2007 νομίζω, Νομίζω ότι αρκετά καλά τα πήγαμε και επίσης η προκήρυξη για υποβολή προσφορών έγινε το 2014 και δεχτήκαμε γύρω στις 400 προσφορές προτάσεις από το αποκρατικό τομέα δημόσιο και από το ιδιωτικό. It, is giving and it should give a big impetus to the European tourism policy because you might have... Οπότε από την ε, Τρίτη όπως ε, παραδοσιακά γίνεται είχαμε αυτή την μεγάλη ισπανική εκδήλωση στη Μαδρίτη και ο Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού επίση δημοσίευσε τα δεδομένα, τα στοιχεία που είχε το 2014 και φτάσαμε σε 457 εκατομμύρια αφήξεων τουριστών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και από τρίτες χώρες. Οπότε το 40% των αφήξεων σε όλο τον κόσμο από το 2010 παρά το ότι όλο ένα και περισσότερο αναδύονται νέοι προορισμοί και είμαστε η δεύτερη περιοχή του κόσμου πλευράς ανάπτυξη σε σχέση με πέρσι και έχουμε επίσης αύξηση 5,3% μόνο η Βόρειος Αμερική μας πέρασε. put in place or years ago for the, on the visa facilitation. Έχουμε επίσης και τα θέματα θεωρήσεων διαβατηρίων Αυτό αφορά επομένω και, τις, ε, και τους αμερικανικούς προορισμούς. Βέβαια δεν είναι αυτός ο καλύτερος μας δείκτης. Θα θέλαμε να έχουμε την ίδια πρόοδο και όσον αφορά την υποδοχή, όσον αφορά μάλλον τι, το πόσο δαπανούν οι τουρίστες. Η αύξηση θα φτάσει το 2% για φέτος. Πάντως ε, δεν πειράζει, έτσι είναι η ζωή. Γιατί ο ανταγωνισμός είναι πάρα πολύ σκληρός. Επίσης, τελευταία τετραετία είχαμε δύο πολύ σημαντικά κοινοτικά νομοθετήματα. Αναθεωρήσαμε την οδηγία την ταξιδιωτική Έγινε η πρώτη ανάγνωση κατά την προηγούμενη θητεία του Κοινοβουλίου. Ίσως ήταν γρήγορη και το Συμβούλιο τον Δεκέμβριο ολοκλήρωσε τη γενική προσέγγιση και η πρώτη συνάντηση τριλόγου τεχνικού θα αρχίσει την επόμενη εβδομάδα. Άρα είναι κρίσιμε οι ώρε, θα πρέπει ακόμα να ξεκαθαρίσουμε κάποια ζητήματα, να βελτιώσουμε την κατάσταση. Οπότε ελπίζω και η δική σα επιτροπή από κοντά να παρακολουθήσει τη εργασίας της Επιτροπής ΣΥΜΚΟ. Και δεύτερο σημαντικό νομοθέτημα ήταν μια άλλη αναθεώρηση που μεγάλη πτυχία προς Κομισιόν η κοινή υιοθέτηση από την Επιτροπή μετά από δουλειά δύο ετών για τα των θεωρήσεων διαβατηρίων του Σέγγεν κυρία Μάλστον και ο κύριος Σταγιάννη τότε είχαν ξεκινήσει τη διαδρομή αυτή. Οπότε και τον Απρίλιο η Επιτροπή ενέκρινε αυτή την αναθεώρηση. Είχαν ολοκληρωθεί συζητήσει στο Κοινοβούλιο και αφορούσε αυτό όλο το πακέτο και είχαμε επίση κυρίω αρμόδια επιτροπή την Λίμπεδα στο Κοινοβούλιο. Θα ασχοληθεί τώρα η καινούργια Λίμπε αυτή τη θητεία την επόμενη εβδομάδα νομίζω. Βέβαια, εδώ έχουμε κάποια κακά μαντάτα, ότι δηλαδή το Συμβούλιο αφήρεσε κάθε μέτρο απλούστευσης, εναρμόνισης το 80-90% δηλαδή των δικών μας προτάσεων. Θα τα ξέρετε γιατί έχουμε επικοινωνήσει επανειλημμένα από το Σεπτέμβριο. Δεν πήγαν καλά οι επαφές με το Συμβουλίο. Άρα θα πρέπει εσείς να καταβάλλετε τιτάνια προσπάθεια για να καταλήξουμε πάλι σε κάτι το οποίο θα βοηθά, θα διευκολύνει τουρισμό και οικονομία. Και να καταλήξετε στους επόμενους μήνες σε κάποια ολοκλήρωση της πρώτης ανάγνωσης, αλλά γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό. Αυτό το 40% των αφήξεων, ιδίως από χώρες που δεν απαιτούν ε, βίζα, να το κρατήσουμε. Αυτά. Έτσι. Επίσης, πετύχαμε να περιλάβουμε στα διορθωτικά ταμεία στην περίοδο του MFF πάνω από 200 προγράμματα και έργα γιατί αντίστοιχες περιοχές κάλυψαν αυτές τις προτάσεις για τον τουρισμό που είχαμε. Και επίση με αυτό ασχολήθηκε το Ταμείο για την Ήπεθρο, το Ταμείο Κοινωνική Συνοχής, Εν πάση τόσο υπήρχε έντονο ενδιαφέρον για το για τον τουρισμό και ακόμη περισσότερο ενδιαφέρθηκαν οι περιφέρειες και αυτό είναι πολύ καλό. Άρα, το 2014 έγινε προπαρασκευαστική δουλειά. Το κάναμε αυτό και με την ευκαιρία της προεκλογικής περίοδου, άρα προλιάναμε το έδαφος για την επόμενη επιτροπή, διαβούλευση για τους πιο ηλικιωμένους, για το μέλλον του τουρισμού. Όλα αυτά δημοσιοποιήθηκαν τον Σεπτέμβριο, τα αποτελέσματα δηλαδή των διαβουλεύσεων. Και ξεκινήσαμε με το Ευρωπαϊκό Φόρο του Τουρισμού, κύριε Κράμερ, που είχατε έρθει. Συνεχίσαμε τις διαβουλεύσεις και με την, ε, με την κυρία Κώστα της Επιτροπής Τουρισμού είχαμε τέσσερις άξονες συζήτησης 1η Σεπτεμβρίου, Ευρωπαϊκή Μέρα Τουρισμού. Ήρθατε εδώ στις Βρυξέλλες και κατόπιν αυτών των διαβουλεύσεων είχαμε αυτές τις μεγάλες συναντήσεις των εμπλεκομένων οπότε η νέα Επίτροπος ήταν καλυμμένη 100% και συμμετέσχει στην εκδήλωση της Μαδρίτης την περασμένη εβδομάδα. Για να σας πω τώρα, έχουμε τις 8 βασικές πρωτοβουλίες που ανακοίνωσε η Επίτροπος. Όλα αυτά θα επαναληφθούν και θα αναπτυχθούν στις 17 και 18 Ενάτου στο Λουξεμβούργο επί Λουξεμβουργιανής τότε Προεδρίας. Αυτές οι βασικές πρωτοβουλίες αφορούν αυτή την ευρύτατη συνένεση του δημόσιου τομέα και του ιδιωτικού τομέα. Έχουμε διάφορες προκλήσεις να αντιμετωπίσουμε γιατί μιλάμε για τον τρίτο οικονομικό κλάδο στην Ένωση. Φοβερή συμβολή στα ΕΦ κλπ. Πρόκειται για έναν ε, επίσης ε, οικονομικό κλάδο που είναι ο πιο ανθεκτικός στην ε, κρίση. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι λείπουν οι προκλήσεις. Δημογραφική εξέλιξη <clears throat> και σε ποσοτικούς και σε ποιοτικούς όρους θέλουμε να έχουμε πιο εξελιγμένες μορφές τουρισμού, πιο απαιτητικές μορφές τουρισμού, καλύτερα προσαρμοσμένες στις ανάγκες των τουριστών. Δεύτερη πρόκληση είναι η ψηφιακή επανάσταση που έχει τροποποιήσει πολλές από τις παραδοσιακές μορφές τουρισμού. Το παραδοσιακό υπόδημα που ακολουθείται είναι μια πολύ μεγάλη πρόκληση. Τρίτη πρόκληση έχει <clears throat> μεγάλη πολυπλοκότητα το ρυθμιστικό πλαίσιο για τον τουρισμό. Όχι τόσο σε ευρωπαϊκό επίπεδο που έχουμε 10-15 το πολύ <clears throat> οδηγίες, αλλά σε εθνικό, περιφερειακό, ακόμα και σε τοπικό επίπεδο υπάρχει ένας κικαιώνας <clears throat> από ρυθμίσεις οι οποίες δεν είναι πάντα συμβατές μεταξύ τους και αυτό δημιουργεί μια κατάσταση η οποία δεν είναι ικανοποιητική. Χρειαζόμαστε λοιπόν όχι μόνο η Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και οι τοπικές και εθνικές αρχές να θέσουν κάποια τάξη σε όλα αυτά. <clears throat> Υπάρχει μια σαφής ανάγκη να αυξήσουμε τις δεξιότητες των εργαζομένων στον τομέα του τουρισμού, γλωσσικές ικανότητες, ικανότητες εξυπηρέτησης και ιδίως για τους τουρίστες που έρχονται από τρίτες χώρες, τα νέα ρεύματα τουριστών από τη Ρωσία, την Ινδία που χρειάζονται διαφορετική αντιμετώπιση. Χρειάζεται λοιπόν να προσαρμοστεί το εργασιακό δυναμικό του τουρισμού στις ανάγκες αυτών των, τουρισμό, τουριστών για να τους παράσχει καλύτερες υπηρεσίες. Χρειαζόμαστε επίσης και πιο υπεύθυνε και βιώσιμες πολιτικές διαχείρισης του τουρισμού. Πρέπει <clears throat> να δείξουμε μεγαλύτερη υπευθυνότητα και εμείς ως τουρίστες όταν ε, ε, μετακινούμαστε μέσα στην Ευρώπη να προστατεύσουμε τους τόπους τουρισμού που αντιμετωπίζουν ήδη προβλήματα. Έχουν γίνει πολλά, αλλά είναι πολλά τα οποία πρέπει να κάνουμε. Επίσης υπάρχει το πρόβλημα της εποχικότητας στον τουρισμό, το οποίο είναι ένα μόνιμο πρόβλημα, το οποίο πρέπει να το αντιμετωπίσουμε και άλλος ένας στόχος είναι να μπορέσουμε να προωθήσουμε καλύτερα τους ευρωπαϊκούς προορισμούς με θεματικά διευρωπαϊκά προϊόντα αυτού του είδους. Να ενισχύσουμε περισσότερο μια θεματική προσέγγιση για τον ευρωπαϊκό τουρισμό. Και θα σας παρουσιάσω τώρα, εν συντομία βέβαια, τις 8 κέρδιες πρωτοβουλίες που, παρουσίασε η κυρία Μπιενκόφσκε. Θα παρουσιάσει λοιπόν την ανακοίνωσή της το καλοκαίρι τις εξής οκτώ πρωτοβουλίες. Καταρχήν, απλοποίηση και ενσωμάτωση της διάστασης του τουρισμού πάντα μέσα στα πλαίσια της επικορικότητας να υπάρξει απλοποίηση του ρυθμιστικού πλαισίου. δεν μπορούμε να παρέμβουμε σε τοπικές και εθνικές ρυθμίσεις, αλλά μπορούμε να ζητήσουμε από τα κρατη να, προ... προχωρήσουν σε μια σοβαρή συζήτηση για το ρυθμιστικό πλαίσιο. Δεύτερον, παράλληλα με την ψηφιακή πρωτοβουλία για την ενιαία αγορά που προετοιμάζουμε, θα πρέπει... Θα πρέπει να βρούμε ένα νέο πλαίσιο οικονομικό, νομικό και κοινωνικό και μια κοινή πλατφόρμα για να μπορέσουμε να συζητήσουμε περισσότερο για την επίπτωση των ψηφιακών εργαλείων στον τουρισμό. Θα προσπαθήσουμε να αποκαλέσουμε αυτή τη συζήτηση. Βέβαια δεν είναι απλό γιατί είναι ένα πολύπλοκο θέμα και είναι ουσιαστικά <clears throat> ένα παγκόσμιο οικονομικό μοντέλο, το μοντέλο των παρόχων ψηφιακών υπηρεσιών με πολύπλοκο νομοθετικό πλαίσιο το οποίο δεν είναι ακόμα επικαιροποιημένο στην Ευρώπη. Αυτή είναι η δεύτερη πρόκληση. Το τρίτο είναι το θέμα της βελτίωσης των δεξιοτήτων. Τέταρτον, να υπάρξει υπεύθυνο και βιώσιμος τουρισμός και να εγκριθεί ο Ευρωπαϊκός Χάρτης για τον υπεύθυνο ε, να εφαρμοστεί μάλλον ο χάρτης για υπεύθυνο τουρισμό και βιώσιμο τουρισμό που ενεκρίθη πριν από δύο χρόνια. Εδώ πρέπει να συμμετάσχουν οι εμπειρογνώμους από τα κρατημέλη, από τις εργατικές ενώσεις, από τον ακαδημαϊκό κόσμο, από την κοινωνία των πολιτών. Θα πρέπει όλοι μαζί να προχωρήσουμε προς την κατεύθυνση αυτή και αυτό πρέπει να γίνει με το καλοκαίρι. <clears throat> Πέμπτη πρόκληση η πρόθεση πρωτοβουλειών που αντιμετωπίζουν το πρόβλημα της εποχικότητας. Θέλουμε να προωθήσουμε πρωτοβουλίες της χαμηλής σεζόν για να μπορέσουμε να καλύψουμε εκεί τα κενά και για τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και για τους Κινέζους που έρχονται από την Κίνα. Υπάρχει ένα σχέδιο λοιπόν ακριβώ για τον τουρισμό από την Κίνα και επίσης συνεργαζόμαστε και με την Βραζιλία και θα εργαστούμε και με τις Ηνωμένες Πολιτείες για να αντιμετωπίσουμε την εποχικότητα έκτη δράση. Και είναι πολύ σημαντικό για την Επιτροπή σας και στον τομέα μεταφορών να εξασφαλίσουμε καλύτερη διαλειτουργικότητα των συγκοινωνιακών μέσων και καλύτερη συνδεσιμότητα των μέσων μεταφοράς, ιδίως για τις περιφερειακές ε, ε, χώρες, για τους προορισμούς που είναι νησιωτικού χαρακτήρα, ε, Έβδομη, η κοινή προώθηση από το δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα όπως, έχει κάνει και, όπως έχουν κάνει οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Αυστραλία, η Γερμανία επίσης με μεγάλους περιφερειακούς προορισμούς. Πρέπει να κάνουμε λοιπόν κάτι τέτοιο να υπάρξει μεγαλύτερη συνεργασία δημοσίου και ιδιωτικού τομέα για την προώθηση του ευρωπαϊκού τουρισμού και των προϊόντων τουρισμού και τέλος και κλείνω εδώ θα προωθήσουμε την καλύτερη διακυβέρνηση στα θέματα τουρισμού. Παντού. Στην Κομισιόν τους τελευταίους τρεις μήνες έχει συνεδριάσει ήδη η Υπηρεσιακή Επιτροπή με τους αρμόδιους επιτροπούς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπάρχει μια σειρά πρωτοβουλειών που ελήφθη και από αυτούς προήλθε και η δημιουργία της ειδική μονάδος Task Force, οι εκθέσεις πρωτοβουλίες, όλα αυτά είναι καλά και χαιρόμαστε πάρα πολύ για αυτές τις πρωτοβουλίες. Θέλουμε επίσης τα κράτη-μέλη να <clears throat> εξασφαλίσουμε ότι θα υπάρξει καλύτερη συνεργασία με τις περιφέρειές τους, να υπάρξει καλύτερη μεταλαμβάδευση πρακτικών και φυσικά θα πρέπει να συνεργαστούμε και με τον ε, τουριστικό τομέα. Δεν υπάρχει ακόμα επαρκή συντονισμός. Θα πρέπει να υπάρξουν καλύτερες πλατφόρμες για τον τομέα τουρισμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να αντιμετωπίσουμε θέματα κοινού ενδιαφέροντος. Αυτό έχει επιπτώσει και στην πολιτική προξενικών θεωρήσεων, πολιτική κοινή προώθησης πολιτιστικών και τουριστικών προϊόντων σε πολλά θέματα κοινού συμφέροντος θα πρέπει ο τουριστικός τομέας να εξασφαλίσει καλύτερη συνεργασία όχι μόνο σε, στο συγκεκριμένο αυτό τομέα αλλά και θέματα που έχουν να κάνουν με τον τομέα της καλλιτεχνικής δημιουργίας, της ε, ένδυσης, της μόδας, ε, ε, του κλάδου υγείας. Θα κλείσω εδώ λοιπόν και είμαι στη διάθεσή σας αν θέλετε να θέσετε ερωτήματα. Στις 3 Σεπτεμβρίου επίσης θέλω να σας υπενθυμίσω έγινε η πρώτη συνάντηση με τον κύριο Φρανσεσκίνη, τον Υπουργό Τουρισμού. Έγινε μια συνάντηση άτυπη των εμπειρογνώμων στον τουρισμό και έχουμε πολλές καλές ιδέες που προήλθαν από αυτή τη συνάντηση. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κύριε Άρτουν. Πρωτού δώσω το λόγο στους συναδέλφους. Θέλω να καλωσορίσω 32 φοιτητές από το Ινστιτούτο Πολιτικών Σπουδών του Μπορντό. Καλώς ήλθατε εδώ και σας δίνω στον κύριο Αντιπρόεδρο αμέσως το λόγο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον κύριο Όρτουν για την παρουσίασή του και πιστεύω <clears throat> χρειαζόμαστε να χρησιμοποιήσουμε περισσότερο χρόνο και να εξετάσουμε όλα αυτά τα θέματα και να μπορέσουμε να αναλύσουμε τις προτάσεις του κυρίου Ορτούν. Ως συντονιστής για την Task Force, την ειδική αυτή δύναμη, μονάδα, <clears throat> σας, ε, ε, ήθελα να σας αναφέρω ότι προφανώς θα αντιμετωπίσω όλα αυτά τα θέματα που αναφέρθηκαν πιστεύω ότι είναι σημαντικό να μπορέσουμε να κάνουμε πιο κατανοητό ότι η έννοια του τουρισμού σημαίνει τουρισμό <clears throat> υπεύθυνο. Υπεστηρίζουμε λοιπόν ιδιαίτερα την ευθύνη στον τομέα του τουρισμού, αλλά φυσικά γνωρίζουμε ότι δεν έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση ιδιαίτερη αρμοδιότητα για αυτά τα θέματα, τα οποία ανήκουν στην αρμοδιότητα των κρατών μελών. Αλλά όπως είπε πολύ σωστά και ο κύριος Όρτου, ο τουρισμός είναι ο τρίτος σημαντικότερος οικονομικός τομέας στην Ευρώπη και πρόκειται για ένα τομέα ο οποίος παίζει σημαντικό ρόλο στην απασχόληση και στην οικονομική ανάπτυξη. Το Κοινοβούλιο λοιπόν και η Κομισιόν Ε, πρέπει να παίξουν κάποιο ρόλο για όλα αυτά και όταν οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου βρίσκονται στις αιστείες τους θα πρέπει να τονίσουν ιδιαίτερα το ρόλο του τουρισμού για την ανάπτυξη των τοπικών αυτών περιοχών. Παρά λοιπόν το γεγονός ότι όπως είπα προηγουμένως δεν έχουμε πραγματικές δικαιοδοσίες και αρμοδιότητες στον τομέα αυτό είναι πάρα πολλά αυτά τα οποία μπορούμε να κάνουμε για να υποστηρίξουμε τον τουριστικό τομέα. μπορούμε να προχωρήσουμε σε άτυπες συζητήσεις μεταξύ μας και να έχουμε σε άτυπο επίπεδο επαφές και διαβουλεύσεις και όπως είπα πέραν της Κομισιόν και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να αντιμετωπίσει το θέμα αυτό. Επομένως, τις επόμενες εβδομάδες και μήνες θα είμαι σε επαφή με την Task Force, την ειδική μονάδα, ώστε να εξασφαλίσω μια μεγαλύτερη ορατότητα αυτού του τομέα και ως μέλος της Επιτροπής Τραν, αλλά και ως μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θέλω λοιπόν να καταθέσω συγκεκριμένες προτάσεις. Νομίζω ότι στην επόμενη ε, συνεδρίαση της ειδική μονάδος θα πρέπει να προσκληθεί και η Επίτροπος κυρία Μπιενκόφσκη. Πρέπει <clears throat> να υπάρχει κάποιο άτομο το οποίο είναι υπεύθυνο για αυτό το τομέα και αυτό το άτομο πρέπει να το προσκαλέσουμε και να έρθουμε σε επαφή μαζί της. Εγώ έχω προτείνει να προσκληθεί η κυρία Μπιανκόφσκη, αλλά στην συνέχεια η συνέλευση των Προέδρων δεν το είχε δεχτεί, γι' αυτό θέλω να επαναλάβω την αίτησή μου στην επόμενη συνεδρίαση της Task Force να προσκληθεί η κυρία Μπιανκόφσκα, γιατί είναι απαραίτητο να μπορέσουμε να προχωρήσουμε σε ένα διάλογο μαζί της. Δεύτερον, έχω κοιτάξει την έκθεση του 2012, 2011 συγγνώμη, που ήταν τελευταία χρονιά που εξεδόθη μια έκθεση για τον τουρισμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση και λαμβάνει υπόψη το νέο νομοθετικό πλαίσιο. Θα ήθελα να ξέρω όμως τι έχει γίνει έκτοτε, τι νέα γεγονότα έχουν λάβει χώρα μετά από το 2011. Όπως ξέρετε είμαι νέος βουλευτής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, παρόλα αυτά με ενδιαφέρει πάρα πολύ αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει ήδη <clears throat> επιληθεί των θεμάτων αυτών πέραν της έκθεσης αυτής και επίσης αν η εκπόνηση αυτής της έκθεσης του 2011 έχει οδηγήσει σε κάποια τα αποτελέσματα. Γι' αυτό θα ήθελα στη δεύτερη συνεδρίαση της Task Force να δούμε ποια ήταν η συνέχεια η οποία δόθηκε στην έκθεση αυτή. Γιατί αλλιώς δεν έχει νόημα να συντάσσουμε εκθέσεις εάν δεν δίνουμε καμία συνέχεια στα πορίσματά τους. Τρίτον, Έχουμε ένα σημαντικό καθήκον. Τις άλλες επιτροπές, την ΛΥΜΠΕ, την ΙΜΚΟ και άλλες που έχουν ε, ενδιαφέρον για τα θέματα του τουρισμού να έρθουμε σε επαφή μαζί τους. Πιστεύω λοιπόν ότι οι περισσότεροι βουλευτές από τις επιτροπές αυτές δεν έχουν αντιληφθεί πλήρως τη σημασία του τουρισμού και είναι δικό μας καθήκον να τους διαφωτίσουμε για τα θέματα αυτά. Θα ήταν χρήσιμο λοιπόν όλοι οι συνάδελφοι και από τις άλλες εμπλεκόμενες επιτροπές να κατανοήσουν το ενδιαφέρον του τουρισμού και εμείς θα πρέπει να τους επιστήσουμε την προσοχή στο θέμα αυτό. Υπάρχουν πολλοί εμπειρογνώμονες οι οποίοι βρίσκονται και εδώ στην αίθουσά μας και υπάρχουν πολλοί ενδιαφερόμενοι φορείς για τα θέματα του τουρισμού και περιμένουν από εμά μέσα στην Επιτροπή Τραν να εξασφαλίσουμε καλύτερη ε, συνέργεια μεταξύ των θεμάτων τουρισμού και των θεμάτων μεταφορών και επιπλέον περιμένουν από εμά να μπορέσουμε να μεταφέρουμε και στους συναδέλφους άλλων επιτροπών την σημασία που επέχει ο τουρισμός. Ελπίζω λοιπόν ότι θα μπορώ να έχω και την υποστήριξη της γραμματείας μας ώστε να γίνουν οι απαραίτητε προσπάθειες και να υπάρξει και η υποστήριξη η οποία απαιτείται για το έργο της Task Force. Έχουμε επίσης την υποχρέωση την ε, εισηγήτρια την Ισαμπέλα Ντελμόντε στην Επιτροπή μας να την υποστηρίξουμε στο έργο της και το είπε και ο κύριος Σορτούν προηγουμένως ότι εδώ έχουμε μια νέα <clears throat> μονάδα, αυτή την Task Force η οποία έχει δημιουργηθεί και η οποία χρειάζεται την απαραίτητη υποστήριξη. Ευτυχώ έχουμε εδώ παρόντα τον επικεφαλής της ε, διαπαραταξιακής ομάδας που ασχολείται με τα θέματα τουρισμού. Θα πρέπει να παραμείνει σε επαφή λοιπόν με την ε, ειδική αυτή μονάδα. Είναι ευρύ αυτή η διαπαραταξιακή ομάδα και ακόμα και αυτοί οι οποίοι δεν είναι μέλη της διαπαραταξιακής ομάδας για τον τουρισμό έχουν τη δυνατότητα να έλθουν σε επαφή με την αρμόδια εισηγήτρια και να τις μεταφέρουν τις προτάσεις τους. Γι' αυτό λοιπόν, ως συντονιστής για το θέμα αυτό, θα ήθελα να εξασφαλίσω την, ε, ότι θα υπάρξει ο απαραίτητος ε, συντονισμός, ότι θα υπάρξει ενδιαφέρον και θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε στον καλύτερο δυνατό τρόπο ε, συνδυασμού του τουρισμού και της των μεταφορών. Θα ήταν κάτι το οποίο θα ήταν ιδιαίτερα αξιέπαινο αν μπορέσουμε να το επιτύχουμε και εγώ θα ήθελα να προτείνω να έχουμε τουλάχιστον μια φορά το μήνα μια συνάντηση της Task Force. Είχαμε πολλές προτάσεις για την ημερήσια διάταξη της ε, Task Force. Θα σας διαβιβάσω αυτές τις προτάσεις και φυσικά με μεγάλη χαρά θα υποδεχτώ περαιτέρω προτάσεις του είδους αυτού και θα ήθελα να παρακαλέσω τον πρόεδρό μας και τη γραμματεία μας στις συνεδριάσεις της Task Force ε, μάλλον στις συνεδριάσεις της Task Force να μην είναι μονάχα ένα σημείο της ημερήσιας διάταξης της Επιτροπής Μεταφορών αλλά να μπορέσουμε να συνεδριάζουμε και ανεξάρτητα από την συνεδρίαση των επιτροπών μας. Να έχουμε λοιπόν μια συνεδρίαση το μήνα <clears throat> της Task Force. Γιατί όταν έρχομαι εδώ δεν είναι εύκολο να βλέπω αμέσως ποιος είναι μέλος της Task Force και δεν ξέρω ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι είναι εδώ για το επόμενο σημείο. Σηκώστε τα χέρια σας παρακαλώ όσοι είσαστε μέλη της Task Force. Ευχαριστώ. Είναι ίσως δύσκολο να έχουμε επικοινωνία μεταξύ μας όταν όλα γίνονται μέσα στη συνεδρίαση της Επιτροπής. Γι' αυτό επαναλαμβάνω την παράκλησή μου να εξασφαλίσουμε ότι θα γίνεται κάπως ανεξάρτητα σε κάποια διαφορετική χρονική στιγμή η συνεδρίαση της Task Force. Αυτό σας το λέω ότι είναι πολύ δύσκολο εάν οι συνεδριάσεις μας είναι εμπεπλεγμένες στην ε, συνεδρίαση της Επιτροπής Μεταφορών και είναι μονάχα ένα σημείο στην γενικότερη ημερήσια διατάξη της Επιτροπής Μεταφορών. Σας λέω και πάλι ότι χαίρομαι για όσα έχει πετύχει η Task Force. Είναι πολύ σημαντικό για μένα να έχω το συντονιστικό ρόλο και πιστεύω και ελπίζω ότι θα συνεχίσουμε να είμαστε πάρα πολύ ενεργοί ως Task Force και θα μπορέσουμε να φέρουμε σε πέρας αυτό το έργο. Θέλω να ευχαριστήσω και πάλι τον κύριο Ορτούν που τόνισε τη σημασία του τουρισμού. Ευχαριστώ κύριε Βέι. Μία διευκρίνηση. Εμείς ως Επιτροπή αποφασίσαμε ότι η Task Force για τον τουρισμό είναι κομμάτι της Επιτροπής μας και αυτό μας εξασφαλίζει και την αίθουσα και τη διερμηνία. Έχουμε 19 μέλη, τα οποία είναι μέλη της Task Force, έχουμε τον κατάλογο στη διάθεσή σας, αλλά αποφασίσαμε όλοι από κοινού ότι οποιοδήποτε ενδιαφέρεται για τα θέματα αυτά θα πρέπει και αυτός να μπορεί να είναι παρόν στις συνεδριάσεις της Task Force. Θέλω να δώσω τώρα το λόγο στον κύριο Φιμ Φαντενκάντ, δύο λεπτά μονάχα γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο. Ε, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν, Εύχομαι καλή επιτυχία στον κύριο Αντιπρόεδρο με την Task Force του για τον τουρισμό. Στην ομάδα μου στο ΕΛΚ οι προσδοκίες μας είναι πολύ ψηλές, πάρα πολύ ψηλές. Και σας εύχομαι πράγματι καλή επιτυχία. Το δεύτερο, Επιτρέψτε μου να χαιρετήσω την παρουσία του Διευθυντή Ορτούνιο τον οποίο και ευχαριστώ για τις πληροφορίες του και τον καλωσορίζω και ελπίζω ότι θα έχουμε έξοχη συνεργασία τα επόμενα 4,5 χρόνια. Πολλοί συνάδελφοι εδώ ενδιαφέρονται για το θέμα αυτό του τουρισμού και θα ήθελα να μιλήσουν και αυτοί. Γι' αυτό θα περιοριστώ σε ένα ερώτημα και μία παρατήρηση. Συμφωνώ με τον Ούγκρο συνάδελφο ότι ο τουρισμός είναι οικονομικός τομέας πάρα πολύ σημαντικός στην Ευρώπη και με τεράστιες δυνατότητες. Όλο και περισσότεροι πλούσιοι από τη Βραζιλία και την Κίνα θέλουν να έρθουν στην Ευρώπη για να διαπράξουν τουρισμό. Ας υποφιληθούμε λοιπόν. Και το ερώτημα τώρα προς τον κύριο Ορτούν είναι τι θα γίνει με το συνδυασμό τουρισμού και ασφαλείας. Λόγω των τελευταίων εξελίξεων, τα γεγονότα των Παρισίων κλπ. Έχουν ληφθεί νέα μέτρα ασφαλείας και χθες ακόμα ελήφθησαν 44 νέα μέτρα από τη Γενική Διεύθυνση Εσωτερικών. Πώς θα συνδυαστούν λοιπόν αυτά τουρισμός και ασφάλεια. Η ασφάλεια είναι ουσιώδης, δεν αμφιβάλλει κανείς, πρέπει να υπάρξει. Πώς όμως θα συνδυαστεί με την ελεύθερη πρόσβαση των τουριστών και τουριστριών κτλ. Κάποτε θα πρέπει να τα συνδυάσουμε. Πώς όμως, πώς νομίζετε κύριε Ορτούν μου ότι θα τα συνδυάσετε και ιδιαίτερα η γενική σας διεύθυνση πώς τοποθετείτε εδώ. Η κυρία Ισαμπέλα Ντελμόντε έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Πρώτα πρώτα πάρα πολύ σωστό το ότι συγκροτήθηκε αυτή η task force, κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, ούτως ώστε να έχουμε κάποιο είδου βοήθεια σε αυτή την πολιτική τουρισμού που είναι τόσο σημαντικό για την Ευρώπη. Γιατί πραγματικά είναι το 10% του ε, εγχωρίου προϊόντο. Και πρόκειται για πάρα πολλού εργαζόμενου σε αυτόν τον κλάδο, ο οποίο δεν μπορεί να θεωρήσουμε ότι είναι ε, ασήμεντο τώρα που βρισκόμαστε σε μια τέτοια συγκυρία κρίση, Οπότε θα πρέπει να στηρίξουμε αυτόν τον τομέα. Οπότε ε, από την Νάπολη να πούμε ότι έχουμε τέσσερα πάνελ και ενδιαφερόμαστε. Έχουμε πάρει μια κατεύθυνση αυτή η πολιτική για, για, για τα ψηφιακά ε, ούτως ώστε να έχουμε κινητικότητα, να έχουμε ενημέρωση ε, και έτσι όλα αυτά να πλαισιώνουν τον τουρισμό. Οπότε θέλουμε να στηρίξουμε μια ευρωπαϊκή πολιτική και να ξεπεράσουμε ε, αυτή την κατάτμιση, την τόσο μεγάλη που υπάρχει ακόμα και σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο και να είμαστε σαν τους ανταγωνιστές μας από τις άλλες υπήρους. Επομένω, να δούμε πώς θα γίνει η ψηφιοποίηση και σε αυτόν τον τομέα, να δούμε πώς θα έχουμε ολοκληρωμένε υποδομές για την ψηφιοποίηση, γιατί στον τουρισμό Πολλέ φορές θεωρούμε ότι είναι χωριστός, ε, ε, χωριστός τομέας, ε, αλλά έχει να κάνει και με την βιομηχανία και με τη γαστρονομία. Άρα θα πρέπει να δούμε πώς θα φροντίσουμε την προστασία του καταναλωτή για την Ευρώπη ως ε, μοναδικό προορισμό, να έχουμε και κάποια οικονομικά μέσα πολιτικής ε, και φυσικά να υπάρχει προσβασιμότητα σε αυτά για να έχουμε ένα βιώσιμο προορισμό. Πέστε μας κύριε Γενικέ, τι σκέφτεστε για την Ευρώπη ως ε, προορισμό. Έχουμε κάποιες αδυναμίες και Πώς βλέπετε ε, τα μέσα πολιτικής που θα μπορούσαμε να ενεργοποιήσουμε για τον τομέα αυτό. Ευχαριστώ. Η κυρία Φώστερ έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Σας κατευχαριστώ πρόεδρε. Και την Κομισιόν για την πολύ συνοπτική της παρουσία, περιεκτική της παρουσίαση, πλήρη. Έχω και εγώ παρελθόν στις ε, αεροπορικές γραμμές και άρα στον τουρισμό και ένα από τα βασικότερα στοιχεία που θέσατε είναι η αξία, η σημασία που έχει για όλες τις χώρες μέλη η οικονομική αξία και για όλους τους τομείς και υπηρεσίες που τον αποτελούν. Είναι μαζική σημασία. Και επίσης δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι υπάρχει τεράστιος ανταγωνισμός στον τουρισμό. Εγώ από το Ηνωμένο Βασίλειο ή κάποιος από την Αυστρία θα χρειαστεί να ανταγωνιστούν οι μεν τους δε, να φέρουν τους επισκέπτες και τους τουρίστες στη χώρα τους. Όλες οι χώρες νομίζω της Ευρώπης έχουν πάρα πολλά τουριστικά προσόντα και δεν είναι έκπληξη που άνθρωποι εκτός Ευρώπης θέλουν τόσο πολύ να έρθουν να την επισκεφτούν. Επομένως, προηγουμένως μπορεί να υπήρχαν όρια και σύνορα και παραπετάσματα, αλλά σήμερα όχι και υπάρχει μεγάλη αύξηση τουριστών και από Αμερική κλπ. Από την Κίνα Ξέρω ότι τα εξετάζετε αυτά τα θέματα των θεωρήσεων, ας πούμε, και της γενικής διευκόλυνσης των μετακινήσεων και του τουρισμού και ότι υπάρχουν εδώ και τίθενται θέματα επικουρικότητας και ασφαλείας. Αλλά θα ήθελα να προσθέσω μερικά θέματα για την τυποποίηση. Πολύ γενικός όρος. Ανέκαθεν λέγαμε ότι θέλουμε να υπάρξουν πρότυπα για την πυρασφάλεια ας πούμε. Ανάλογα με το ξενοδοχείο στο οποίο θα πάτε αν είναι στην Ιταλία ή στη Γερμανία βλέπετε ότι υπάρχουν ομοιότητες ως προς τις κανονισμούς για την πυρασφάλεια. Αυτά είναι όλα πολύ χρήσιμα και πολύ σημαντικά. Καλό είναι λοιπόν που υπάρχει αυτή η Task Force. Θα ήθελα τώρα να σας συστήσω ένα νέο μέλος των συντηρητικών, εδώ που δείχνω. Αλλά πάντως σας ευχαριστώ για την παρουσίασή σας. Μερσή λέει ο πρώτος. Η κυρία Ζέσκου Μπιλμπάου έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Ορτούν για την παρουσίαση που μας έκανε και επίσης να τον ευχαριστήσω για την τοποθέτησή του που ήταν πάρα την ε, κυρία Επίτροπο μάλλον για την τοποθέτησή της που είναι πολύ σαφής. Για τα 8 σημεία πρωτοβουλίας που μας παρουσίασε ο κύριος Ορτούνο σημεία εργασίας μπορούμε πιστεύω να κάνουμε τις απαραίτητες προσπάθειες πρώτα απ' όλα για να έχουμε σαφή ηγετική, ε, ηγετικό ρόλο Δεύτερον, να διευκρινίσουμε καλύτερα του στόχου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε συνεργασία με το Συμβούλιο και την Κομισιόν και να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε ότι θα υπάρχουν οι απαραίτητοι πόροι. Ο κύριο Σόρτουν ανέφερε τι 8 πρωτοβουλίε, τι κέρυε πρωτοβουλίε που θέλει να παρουσιάσει η κυρία Επίτροπο. Επίτροπος τόνισε την ανάγκη βιώσιμου και υπεύθυνου τουρισμού. Εγώ θα ήθελα να θέσω το ερώτημα αν μέσα σε αυτό συμπεριλαμβάνεται και η έννοια του τουρισμού ο οποίο έχει χαρακτήρα είναι ενωτικό Γιατί θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και περιεκτικό τουρισμό. Τα άτομα τα οποία έχουν αναπηρίες και προβλήματα θα πρέπει να δώσουμε τη δυνατότητα να περιληφθούν και αυτοί στην τουριστική δραστηριότητα και να εξασφαλίσουμε τι θέσει εργασία που μπορούν να προέλθουν από αυτό. Πιστεύω ότι υπάρχει και ένα άλλο σημαντικό μήνυμα για την Επιτροπή μα και τα κατημέλη. Μιλάμε για την αύξηση που θα υπάρξει στον τουρισμό μέχρι το 2020-2030. Μιλάμε για την διαλειτουργικότητα των μεταφορών και των τουριστικών υποδομών. Είναι απαραίτητο λοιπόν να δημιουργήσουμε την απαραίτητη αυτή διαλειτουργικότητα μεταξύ των μέσων μεταφορών που πολλές φορές υπάρχουν πολλά προβλήματα όπως φαίνεται από τις εκθέσεις που έχουμε. Έχουμε τους ενιαίους εθέρες, έχουμε το πακέτο για τα λιμάνια, την ψηφιακή ένωση, είναι πάρα πολλά πράγματα λοιπόν τα οποία πρέπει να φέρουμε σε πέρας και τέλος θα ήθελα να πω ότι πρέπει να βρούμε την κατάλληλη αντιμετώπιση για τα θέματα αυτά και στην χώρα των Βάσκων εμείς έχουμε δημιουργήσει ένα επιγραμμικό εργαλείο το οποίο ε, παρουσιάζει την στρατηγική της περιοχής και 75% των τουριστών που έρχονται στην περιοχή της χώρας των Βάσκων κάνουν τις κρατήσεις τους από το διαδίκτυο. Πρέπει λοιπόν να εξασφαλίσουμε τις βέλτιστες πρακτικές σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να μπορούμε όλοι να έχουμε ένα καλύτερο εργαλείο το οποίο θα παρουσιάζει τις προστάσεις στον τουριστικό τομέα. Πρέπει να παίξουμε ηγετικό ρόλο, πρέπει να καθορίσουμε τους στόχους μας και να δώσουμε τους απαραίτητους πόρους και τέλος θα πρέπει να συμμετάσχουν πολύ περισσότερο οι περιφερειακές αρχές που όπως τόνισε ο κ. Σορτούν, αυτές θα πρέπει να βοηθήσουν να καθοριστούν τα νέα σχέδια του μέλλοντος. Ευχαριστώ, λέει και ο πρόεδρος, ο, η Jill Evans. Ευχαριστώ, πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να καλωσορίσω τη σύσταση αυτής της Task Force και να ευχαριστήσω τον κύριο Ρτούν για την παρουσίασή του που κάλυψε πολλές από τις πτυχές του τουρισμού και της τουριστικής πολιτικής. Χαίρομαι που το συζητάμε σήμερα διότι όπως είπαν και άλλοι, υπάρχει εδώ η δυνατότητα οικονομικής ανάπτυξης σε όλα τα τμήματα της Ένωσης. Έχει πολύ μεγάλες δυνατότητες που δεν τις έχουμε ακόμη εκμεταλλευτεί. Η βιώσιμη ανάπτυξη μέσω του βιώσιμου τουρισμού εξαρτάται από πολλούς άλλους παράγοντες φυσικά όπως τις καλές μεταφορές και συγκοινωνίες με πολιτιστικά, βιομηχανική, θέμα τοποθεσίες βιομηχανικής κληρονομιάς κλπ. Επίσης, έγινε λόγος εδώ για κοινοπραξίες ιδιωτικού δημόσιου τομέα, αλλά θα ήθελα συγκεκριμένα να μιλήσω για το ρόλο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που είναι βασικοί παράγοντες εδώ, ιδίως σε περιφερειακό επίπεδο και που έχει όλο και μεγαλύτερη σημασία. Τι προτείνει λοιπόν η Κομισιόν ειδικά για την στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στον τουρισμό. Η κυρία Αγιάλα Σέντερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Ορτούν που ήρθατε και μας ε, τα είπατε τόσο με το τέτοια πληρότητα και ε, εις βάθος. Ε, φαντάζομαι ότι αυτό αποδεικνύει το πόσο έχετε πάρει στα σοβαρά την υπόθεση του να δοθεί μια όθηση σε αυτόν τον τομέα που τόσο πολύ ε, έχει πληγεί και από την κρίση και είναι τόσο ευάλωτος και επίσης έχει πληγεί από την ε, υπόθεση της σύγκρουσης της Ρωσίας με την Ουκρανία. Και στην Ισπανία έχουμε πληγή όσον αφορά ακριβώ το ότι ο τομέα αυτό είναι ευάλωτο. Γίνονται με διάφορε κρίσει, ε, πλήσεται η Ευρώπη και α μην είναι αυτή στη, στη ρίζα, στην αιτία των ε, κρίσεων και των συγκρούσεων. Άρα θα πρέπει να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για να αντιδράσουμε. Και υπάρχει επομένω κάτι άλλο βασικό και ιστορική σημασία. Το τι γίνεται με τι θεωρήσει των διαβατηρίων. Αυτό δεν είναι δικό μα είναι θέμα τη επιτρο... δική μα επιτροπή, είναι θέμα άλλων επιτροπών. Όμω είναι θέμα το οποίο έχει μεγάλη σημασία ε, για τους τουρίστες από Βραζιλία, Φερρυπίν, ε, η Κίνα. Ε, υπάρχουν πάρα πολλοί. Να, και από την άλλη μεριά Μεσογείου συνέχεια ανακύπτει αυτό το θέμα. Βέβαια έχει ασχοληθεί ο κύριος Σταγιάννη. Τι γίνεται τώρα όσον αφορά τον προϋπολογισμό. Πάντα εκεί υπήρχε κάποια απογοήτευση σε σχέση με την προηγούμενη θητεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής γιατί τελικά δεν είναι το ίδιο όπως σε άλλους τομείς ούτως ώστε να μπορέσει να πρικοδοτήσει η Κομισιόν αυτόν τον τομέα. Έλειπε μια νομική βάση που να εκάλυπτε 100%. Εγώ νομίζω ότι με αυτά που έχουμε στα χέρια μας μπορούμε να δουλέψουμε. Εν πάση περιπτώσει, αν υπάρχει μια τέτοια νομική πλαισίωση, να πρέπει να δούμε κύριε Ορτούνου μήπως τελικά το καταφέρουμε στα επόμενα χρόνια. Δεν, δεν αργώ άλλο πρόεδρε και θέλω να σας ξεκαθαρίσω ότι η Task Force, εμείς που δεν συμμετέχουμε, παρόλα αυτά ενδιαφερόμαστε. Αυτή η Task Force, όπως λέγαμε πάντα, είναι ανοιχτή σε όλους. 19 είναι τα μέλη της. Δεν είναι πάρα πολλά τα μέλη τα σημερινά, το οποίο τώρα συμμετέχουν αλλά θα πρέπει να δούμε το πώς και έτσι επίσημα θα βοηθήσουμε τον τουρισμό. Η Task Force είναι ένα βήμα πρόοδο. Σας παρακαλώ να κρατήσετε το χρόνο ομιλίας για να μην εμποδίσετε του άλλους να λάβουν το λόγο. Ο κύριος Δε Καντε Πασκάλ. Ναι. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Ορτούν για την παρέμβασή σας. Νομίζω ότι οι οκτώ προτάσεις που αναφέρθηκαν από την πλευρά της αρμοδίας επιτρόπου είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσες. Θα, θα πρέπει να μπορέσουμε να τις ε, ε, αντιμετωπίσουμε. Ξέρω ότι ο πρόεδρος ε, δεν μου επιτρέπει να μιλήσω για πολύ χρόνο, αλλά υπάρχει ένα θέμα που εγώ ως Ισπανός δεν μπορώ να το παρακάμψω και είμαι αντιπρόεδρος αυτής της ε, διαπαραταξιακής ομάδας για τον τουρισμό για μας που είμαστε η τρίτη μεγαλύτερη τουριστική δύναμη μετά, στον κόσμο μετά τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Γαλλία. Είναι κέριος ο τουρισμός. Έχουμε μεγάλη εμπειρία στο θέμα αυτό και θέλουμε να υπάρξει μεταλαμβάνευση βελτίστων πρακτικών και επίσης να αναφέρουμε και τις κακές πρακτικές που θα πρέπει να διορθωθούν. Συμφωνώ με το πνεύμα αυτής της πρωτοβουλία για λιγότερη και καλύτερη ρυθμίση και νομοθεσία. Πρέπει να χρησιμοποιήσουμε λοιπόν την ε, ε δημιουργικότητά μας γιατί έχουμε το άρθρο 95, το 55 συγγνώμη για την εναρμόνιση, που δεν μας δίδει πολλές δυνατότητε για τις βέλτιστες πρακτικές. Αυτή τη στιγμή η Ισπανία ενδιαφέρεται ιδιαίτερα να αγωνιστεί και αυτή κατά της εποχικότητας, να βοηθήσει τον τουρισμό των νέων και της τρίτης ηλικίας και να δώσουμε μεγαλύτερη έμφαση στην ποιότητα και όχι στην ποσότητα στον τουρισμό. Θέλουμε λοιπόν να τονίσουμε ότι είναι πάρα πολλοί από τους νέους που έρχονται με το Εράσμους στην ε, Ισπανία. Προτιμούμε να είναι πραγματικά τουρίστες και όχι άτομα τα οποία έρχονται εδώ στην Ισπανία μόνο για τον ήλιο και για να πιούν. Θέλουμε λοιπόν να έχουμε ένα τουρισμό υγείας, ένα τουρισμό τρίτη ηλικία, όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά και είναι απαραίτητο να έχουμε μεγαλύτερη επαφή σε πολιτιστικό επίπεδο, όπω είπε η κυρία Μπιλμπάου, να είναι περιεκτικό ο τουρισμό και να μπορεί να βοηθάει και το πολιτιστικό πλαίσιο. Θέλω να ευχηθώ κάθε επιτυχία λοιπόν στην Task Force και ελπίζω θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε όλοι από κοινό. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ. Θέλω να κάνω ένα σχόλιο σύντομα. Καταρχήν το θέμα των περιφερειών. Είπε δικαίως και η Κομισιόν ότι στα περιφερειακά προγράμματα στο σύνολο της Ευρώπης είναι πάνω από 200, περιλαμβάνεται μια στρατηγική και για, το στρατηγική και για τον τουρισμό. Άρα μεγάλο τμήμα του... των χρημάτων που δίνουμε για τον τουρισμό περνάνε από το Περιφερειακό Ταμείο. Αυτά τα ξέρω, ήμουν και στην Επιτροπή των Περιφερειών και ξέρω ότι από αυτό το ταμείο δίνονται τα χρήματα. Εξού και μία συμβουλή που θέλω να δώσω στην Task Force. Να συνεργάζεστε με τη Γενική Διεύθυνση Περιφερειών για την Περιφερειακή Ανάπτυξη και τον Τουρισμό. Τώρα για την καινοτομία είναι κάτι που λείπει εδώ η Ευρώπη, στην Ευρώπη. Εγώ είμαι από μια περιφέρεια που έχουμε ειδικευτεί στα χειμερινά σπορ. Πριν από 10 χρόνια κάναμε πολλές καινοτομίες συνδυασμού αθλητισμού με τουρισμό και διασκέδαση και με πολλές νέες εγκαταστάσεις. Άρα ο τουρισμός μπορεί να οθήσει και άλλους τομείς και άλλες δραστηριότητες παράπλευρες. Πρέπει λοιπόν να τονίσουμε περισσότερο το θέμα της καινοτομίας, όπου ο τουρισμός μπορεί επίσης να παίξει ένα ρόλο. Και πρέπει να τα δούμε όλα αυτά, να δούμε τι υπάρχει στην Ευρώπη και τι λείπει. Κλούν. Ήταν ενδιαφέρουσα αυτή η παρουσίαση του κυρίου Ορτούν και είναι πολλά θέματα τα οποία ενδιαφέρουν τις επιχειρήσεις και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ιδίω για να υπάρξει απλοποίηση των διατάξεων, καλύτερη βελτίωση των προσόντων των εργαζομένων. Νομίζω ότι μια τέτοια ειδική μονάδα θα πρέπει να είναι πιο συγκεκριμένη σε αυτά τα οποία θα την απασχολήσουν. Όλοι αυτοί οι οποίοι παρέχουν τουριστικά προϊόντα θα πρέπει να εξασφαλίσουν ότι θα βελτιώνουν τις δεξιότητές τους, θα αναπτύσσουν ένα καλό προϊόν. Και από τη δική μας πλευρά θα πρέπει να τονίσουμε την προσβασιμότητα, <clears throat> τις καλύτερες μεταφορικές συνδέσεις. Έρχομαι από μια νησιωτική περιοχή της Ιρλανδίας και υπάρχει μεγάλος ανταγωνισμός με άλλες περιφέρειες είναι πάρα πολύ σημαντική η εξασφάλιση μεταφορικών συνδέσεων με την ε, Ιλανδία. Εσείς υποστηρίζετε τα τρένα, αλλά εμεί τι να τα κάνουμε τα τρένα. Εκεί χρειαζόμαστε να έχουμε περιφερειακά αεροδρόμια, είναι πάρα πολύ σημαντικά. Όλα αυτά λοιπόν πρέπει να είναι τμήμα της αντιμετώπισης για κάθε μία από τις 200 περιφέρειες της Ευρώπης και πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να υποστηρίξουμε οποιαδήποτε σύνδεση υπάρχει σε κάθε περιφέρεια, στη συγκεκριμένη περίπτωσή μα τα περιφερειακά αεροδρόμια, γιατί αλλιώ δεν μπορούν να έρθουν οι τουρίστες στην περιοχή μας και όπως είπε και ο κύριο Ορτούν, είναι απαραίτητο να εξασφαλίσουμε την ανάπτυξη αυτών των περιοχών. Ευχαριστώ. Η Κλάουδια Νίλα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι εδώ συζητούμε ένα θέμα το οποίο είναι σημαντικό και κέριο, το θέμα του τουρισμού. Είναι μια πάρα πολύ σημαντική οικονομική δραστηριότητα ο τουρισμός και είναι συγχρόνως αποφασιστικός ο ρόλος του τουρισμού για την ανάπτυξη των περιοχών μας. Κάποιες περιοχές είναι περιοχές οι οποίες είναι απομεμακρυσμένες και απομονωμένες, αλλά είναι πολύ σημαντικό ε, να αναπτύξουν τον τουρισμό και αυτό αφορά ιδίως την περιοχή από την οποία προέρχομαι, την Μαδέιρα. Είναι πολλές οι δυνατότητες για να αναπτυχθεί ο τομέας του τουρισμού εκεί. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Ορτούν, τον Γενικό Διευθυντή που παρουσίασε το πρόγραμμα της Κομισιόν και θα ήθελα να υπογραμμίσω και ένα σημείο το οποίο για μένα είναι θεμελιώδες. Είδες αναφέρθηκε αυτό το θέμα της ανθεκτικότητας των επιχειρήσεων. Όταν όλη η Ευρώπη περνάει μια μεγάλη οικονομική κρίση, ιδίω σε ορισμένα κράτη-μέλη, υπήρξε μια πολύ μεγάλη ένταση της πίεσης της επιχείρησης. Θα ήθελα να θέσω και το εξή ερώτημα. Σε επίπεδο χρηματοδότησης, ποια είναι η πρόθεση της Κομισιόν <clears throat> και πώς θα μπορέσει να βοηθήσει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις για να παίξουν το ρόλο αυτό που απαιτείται από αυτές. Και επίσης ό,τι αφορά την περιφερειακή διάσταση και προερχόμενη από τη Μαδέιρα, θα ήθελα να ζητήσω πώς βλέπει η Κομισιόν το θέμα των συμπλεγμάτων, των clusters, σε, σε ό,τι αφορά τον τουρισμό ε, των παρακτήων περιοχών. Πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν να αντιμετωπίσουμε τα θέματα αυτά των περιφερειακών αεροδρομίων που ανέφερε και η προηγούμενη ομιλήτρια και την καλύτερη προσβασιμότητα μέσω εναερίων συγκοινωνιών. Ευχαριστώ πολύ. Η Ελίζαμπεθ Ρόζενμπεργκ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ε, αναμφίβολα ο τουρισμός στην Ευρώπη σε επίπεδο ανταγωνισμού αντιμετωπίζει προβλήματα σε σχέση με τις άλλες υπήρους, αλλά παρά κατά την άποψή μου, κατέχει τα πρωτεία. Εμείς όταν είχαμε την ελληνική προεδρία η Ελλάδα προώθησε πάρα πολύ το θέμα του ευρωπαϊκού τουρισμού με διεθνή συνέδρια, με συνέδρια υπουργών όπως ξέρετε και η χώρα μου παρά το γεγονός ότι βρίσκεται σε βαθιά κρίση φέτος είχε εξαιρετικά, εξαιρετικές επιδόσεις στο θέμα του τουρισμού. Όμως το θέμα του εποχικού τουρισμού το οποίο ανεδείχθη από τον ε, κύριο Ορτούν και τον ευχαριστούμε πολύ για τη σημερινή αναλυτική του εξιστόρηση και των οκτώ σημείων της Ευρωπαϊκής της ε, Επιτρόπου ε, συγκρούεται διότι στις άλλες υπήρους περίπου δεν υπάρχει εποχικός τουρισμός, υπάρχει διαχρονικός τουρισμός. Εδώ, ενώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση το παρατηρούμε από χώρα σε χώρα, το φαινόμενο να παρατηρείται. Ε, προσωπικά σας ευχαριστώ που μετέχω στην Task Force. Θεωρώ ότι ήταν πολύ σημαντικές οι παρατηρήσεις που έγιναν από τον κύριο Wayne, τον συντονιστή, σε σχέση με την δραστηριότητα που μπορεί να έχει η Task Force παρά τις πολύ περιορισμένες δυνατότητες που έχει η Επιτροπή μας στον ευρύτερο τομέα αυτό. Ε, ε, πήρα το λόγο γιατί ήθελα να ρωτήσω ειδικά την Επιτροπή, κύριε Πρόεδρε, κατά πόσον έχει γίνει μια αναλυτική παρατήρηση των αδυναμιών που υπάρχουν σε σχέση με τον ανταγωνισμό στον ευρωπαϊκό τουρισμό συγκριτικά με τον διεθνή τουρισμό, δηλαδή με τον τουρισμό στις άλλες υπήρους. Σας το λέω γιατί παράδειγμα χάρη εμείς ε, στη χώρα μου αντιμετωπίσαμε προβλήματα με τα γεγονότα στην νοτιοανατολική Μεσόγειο από την γείτονα Τουρκία η οποία έχει τουριστικό προϊόν και μπορεί να μας ανταγωνιστεί και ήταν άνισος ο τρόπος εννοώ. Και η δεύτερη ερώτηση που ήθελα είναι αν γίνονται σκέψεις από την Επιτροπή για μια ενισχυμένη η οικονομική ενίσχυση των χωρών που βρίσκονται σε κρίση. Προσωπικά ξέρετε ότι πια είναι πολύ λίγες, αλλά η χώρα μου βρίσκεται σε πρόγραμμα και έχει πληγεί ως προς τις υπηρεσίες του τουρισμού οικονομικά. Αν υπάρχει δηλαδή πρόβλεψη για μια ενίσχυση πάνω σε αυτό το τομέα, και κλείνοντας θα ήθελα να συμφωνήσω με τον συντονιστή της Task Force όχι κατά ανάγκη για ιδιαίτερες ε, ε, συναντήσεις της Task Force μέσα εκτός του πλαισίου της Επιτροπής μας, αλλά πιο συχνές που μπορεί να γίνονται και σε ένα πιο περιορισμένο επίπεδο και ο καθένας από τη χώρα του, αλλά και από την πολιτική του ομάδα να εισφέρει πληροφορίες που θα είναι κρίσιμες στην εργασία από κοινού που γίνεται. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ. Ε, για την κυρία Κλούνη θέλω να πω ότι με, είπατε ότι είμαι μανιακός για τα τρένα αλλά καταλαβαίνω δεν μπορεί να γίνει αυτό σε όλα τα νησιά και το κάνω αυτό λαμβάνοντας ο ίδιος το λόγο. Πιστεύω ότι μπορούμε να υποστηρίξουμε γενικά τις συνδέσεις για τι περιφερειακές περιοχέ. Όταν έχουμε περιοχέ οι οποίε είναι μακρινέ, αυτό έχει νόημα. Αλλά Τώρα το να υποστηρίξουμε όλα τα περιφερειακά αεροδρόμια τα οποία στη χώρα μου έχουν χρεοκοπήσει τα περισσότερα, αυτό δεν έχει κανένα νόημα. Θέλουμε να εξασφαλίσουμε την κινητικότητα, αλλά για περιοχές οι οποίες πραγματικά δεν έχουν άλλες δυνατότητες. Είπατε επίσης, κύριε Ορτούν, ότι σε ορισμένε περιοχές στην ε, Γερμανία, στην Φιλανδία και στην ε, Σουηδία μπορεί κανείς να κάνει θαυμάσιες εκδρομές, ακόμα και το χειμώνα, με το ποδήλατο και στην Αυστρία. Μπορούμε λοιπόν με αυτόν τον τρόπο να προωθήσουμε τον τουρισμό και μπορούμε να τονίσουμε ότι ο τουρισμός ποδηλατικού χαρακτήρα έχει αυξηθεί με ρυθμούς 20% το χρόνο. Είναι καλύτερα να πηγαίνει κανείς με ποδήλατο παρά με ε, αυτοκίνητο. Με απλές υποδομές μπορούμε να έχουμε πολλά πλεονεκτήματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο δεν χρειάζεται λοιπόν το κόστο το οποίο χρειάζεται για του αυτοκινητοδρόμου και είναι εξάλλου και πολύ καλό και για την υγεία. Δεν είναι <clears throat> τυχαίο ότι οι ποδηλάτε ζουν πέντε χρόνια περισσότερο κατά μέσον όρο από του μη ποδηλάτε. Και φθηνά είναι και ευχάριστα είναι και υγιεινά είναι. Επομένω, ο ποδηλατικό τουρισμό είναι ο τουρισμό του μέλλοντο. Ξαναδίνω λοιπόν το λόγο στον κύριο Ορτούν. Thank Σας ευχαριστώ πολύ όλους, όλους για τα καλά σας λόγια, την υποστήριξη, τις προτάσεις σας. Από ό,τι κατάλαβα έχουμε μέχρι 10 και μισή, αλλά θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος και να μην παραλείψω να απαντήσω σε κανέναν, ε. να απαντήσω σε όλα όσα είπατε και σχολιάσατε. Καμιά φορά βέβαια δεν είναι τόσο εύκολο. Αρχίζω φαντικά ξεκίνησε με εύκολη ερώτηση. Πώς να εξισορροπήσουμε ασφάλεια με τουρισμό. Να σας πω. πρώτο πρώτο, Προσωπική άποψη. Γιατί δεν είναι βέβαια η ασφάλεια δική μου αρμοδιότητα. Η κυρία Μογκερίνη και άλλοι συνάδελφοι ασχολούνται με αυτά. Εμείς από την οπτική γωνία του τουρισμού. Θεωρούμε ότι και για τους τουρίστες είναι σημαντική υπόθεση η ασφάλεια. Από κάποιες τρίτες χώρες είχαμε καταγγελίες για έλλειψη ασφάλειας. Όχι όμως ε, με την έννοια της τρομοκρατίας. είχαμε πρόβλημα με επίθεση κατά κάποιων ε, Κινέζων τουριστών ε, για να τους κλέψουν κάποια ε, αντικείμενα πολυτελείας κλπ. Άρα για την πολιτική του τουρισμού είναι σημαντικό και άρα αυτό θα πρέπει να τα κράτη-μέλη. Και αυτό δεν αφορά μόνο τους πολίτες τρίτων χωρών, αλλά αφορά και τους Ευρωπαίους να είναι δηλαδή οι πόλεις ασφαλέστερες. Τι να σας πω, θυμάμαι ε, τι γινόταν με τον κύριο Ταγιάννη. Λέμε ότι αν θέλουμε να συνδέσουμε ε, την αναθεώρηση της ε, πολιτικής για τις βίζες των διαβατηρίων με την ασφάλεια. Ε, τότε εδώ πέρα αυτό δεν είναι το πιο σωστό γιατί είπαμε τι γίνεται με την τρομοκρατία. Είναι θέμα το οποίο έχει βγει τώρα τις τελευταίες 15 μέρες. Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί η πολιτική τη θεώρηση διαβατηρίων ούτω ώστε να αντιμετωπίσει κανεί του ε, τρομοκράτε που έρχονται από το εξωτερικό. Γιατί πάρα πολύ συχνά ήδη βρίσκονται στα κράτη-μέλη ε, οι τρομοκράτε. Άρα δεν πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τι βίζε για τέτοιου είδου ασφάλεια. Τώρα, έχουμε θέματα ε, καθαρά ασφαλείας. Είναι θέμα κρατών μελών, το συντονίσουν τους ε, διασυνοριακούς ελέγχους και πολιτική μετάσταση βεβαίως σχετίζεται με τον τουρισμό αλλά ε, κατά τη γνώμη μας όχι δεν θα θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε για ασφάλεια την πολιτική των θεωρήσεων. Έχουμε την ε, ε πολιτική, την εξωτερική μας πολιτική, έχουμε, έχουμε άλλα, άλλους τρόπους. Τώρα, η κυρία Ντεμόντε. Αυτό που σας ενδιέφερε ήταν το ότι χρειάζεται καλύτερη προώθηση, διαφήμιση της Ευρώπης. Για όλους αυτούς τους προορισμούς που έχουμε εδώ, είναι φυσικά και έχουμε η πιο πλούσια ήπειρος από πλευράς ε, κληρονομιάς, ε, από πλευρά ποικιλία, ε, πολιτιστικά, ε, φυσικό περιβάλλον, ε, όλα αυτά τα μνημεία. Άρα αυτό θα πρέπει να γίνει ανταγωνιστικά. Μάλλον συγγνώμη, πρέπει να γίνει με συνεργασία και όχι με ανταγωνισμό μεταξύ των κρατών μελών. Βεβαίω να έχουμε εδώ συνεργασία κρατών μελών. Πολλά μπορεί να γίνουν και να φέρουν και οικονομία κλίμακας. να έχουμε διακρατικές εκστρατείες διεθνιστικές. Έχουμε, είπαμε, Ρώσους, Αμερικάνους, Βραζιλιάνους που ενδιαφέρονται και αν έχουμε κάποια προϊόντα ελκυστικά για εκείνους, ε, τότε αυτοί έρχονται στην Ευρώπη. Στο Λονδίνο, στη Βενετία. Τέλος πάντων έρχονται στην Ευρώπη. Άρα θα πρέπει ε, συνδυάσουμε τους οργανισμούς τουρισμού, τις περιφερειακές αρχές και έτσι όλοι μαζί να διαφημίσουμε τους προορισμούς της Ευρώπης. Γελία είναι η πρικοδότηση βέβαια που έχουμε γιατί θα πρέπει να σας θυμίσω ότι το άθροισμα των προϋπολογισμών για τους εθνικούς οργανισμούς τουρισμού πάνε περίπου, περίπου στα, στο ένα εκατομμύριο ευρώ. Ένα δις, ένα δις. Και σορτούν. Αλλά από, σε σχέση με τον, με προπολογισμό αυτό, σε σχέση με αυτό λοιπόν δίνουμε μόνο μόλις ένα εκατομμύριο για ε, διαφήμιση. 90 εκατομμύρια δίνουν οι Ελβετοί. Οι Γερμανοί που έχουν τόσους προορισμούς, Βαβαρία, Βερολίνο, Ρήνο, 60 εκατομμύρια ευρώ. Βλέπετε τι γίνεται. Άρα θα πρέπει να διαθέσουμε περισσότερα χρήματα. We have a lot to do. We will put these things on the table. Πρέπει επομένω να δούμε πώ θα έχουμε περισσότερα χρήματα που θα διαθέσουμε να συνεργαστούμε και ελπίζω ότι σε μια διετία θα έχουμε έτοιμη μια καινούργια πρωτοβουλία τώρα. Προσωποποίηση. Είπατε για το θέμα της πυρασφαλείας, παλιά ιστορία αυτή, συστάσεις έχουμε της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το 86 επικαιροποιήθηκε, ε, άλλαξε. Ακόμα και υπάρχουν πολλά που πρέπει να γίνουν και σε αυτόν τον τομέα. Εδώ δεν χωράει εναρμόνιση, αυτό είναι πρόβλημα, αλλά μπορούμε να κάνουμε περισσότερο. Ο κύριος Τίμερμανς είπε για καινούργια νομοθεσία, σοβαρές προτάσεις και κάποιες πρωτοβουλίες οι οποίες να είναι δυνατόν να τις παρακολουθούμε, να τις δοκιμάζουμε, να έχουν διαφάνεια. Ακόμα δεν φτάσαμε εκεί που θα έπρεπε και οι περιφέρειες βέβαια έχουν στα χέρια τους πάνω από τη μισή νομοθεσία. Και συνεργαζόμαστε, έχουμε τα δίκτυα έχουμε τα κλάστερς αυτούς τους κόμβους για συνεργασία με τις περιφέρειες. Έχουμε αυτό το δίκτυο ευρωπαϊκών επιχειρήσεων. Και υπάρχει και η διάσταση μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Και φυσικά ο καλύτερος τρόπος είναι μέσω των περιφερειακών πρωτοβουλειών. Ψηφιακά, Έχουμε αυτό το πόρταλ για τις ΜΜΕ, αυτή τη διαδικτυακή πύλη και είπαμε το καλύτερο είναι να ασχοληθούμε σε περιφερειακό επίπεδο. Η Νένς έχεις δίκιο, έχουμε αυξήσει την ε, πρικοδότηση 2-3 εκατομμύρια τα τελευταία χρόνια έχουμε προσθέσει. Πάμε για 10, 12 με, με τις προπαρασκευαστικές δράσεις. Φτάνουμε στα 15 εκατομμύρια. Αν ρίξετε μια ματιά στον προπολογισμό και του 16, είδατε τι έγινε γύρω στα γένεια. 105 εκατομμύρια τα τελευταία 5-6 χρόνια. Και στο προσωπικό είχαμε, ήμασταν 15 το 2010 και τώρα είμαστε 24. Δεν είναι τόσο άσχημη κατάσταση. Αν έχουν προσωπικό 24 αξιόλογων στελεγών που κάνουμε πολλά. Ναι, τι γίνεται τώρα με, με, με την ε, νεκρή τέλο πάντων περίοδο που δεν είναι περίοδο αιχμής. 128 προτάσεις είχαμε όταν κάναμε αυτή την πρόσκληση υποβολή προσφορών για νέου, για ηλικιωμένου. Δηλαδή τα διπλάσια από ό,τι τα αναλύσαμε όλα αυτά και θα πρέπει να δούμε τι γίνεται από πλευρά ποιότητα, από πλευρά συνεργασία, ε, συγκρατικού τομέα, ιδιωτικού τομέα. Ένα άλλο τώρα θέμα. Προσβασιμότητα. Τι άλλο ρωτήσατε. Ποιος το είπε. Α, η κυρία Μπιλμπάου. Ναι, ναι, βεβαίω και θα με αυτό. Πάρα πολλές προτάσεις για προσβάσιμο τουρισμό. Η προσβασιμότητα είναι αναπόσπαστο τμήμα της έννοιας του υπεύθυνου τουρισμού βεβαίω. Και θα έχουμε και τον χάρτη του ευρωπαϊκού τουρισμού. Θα δείτε. Νομίζω ότι απάντησε σε όλα. Α, για τις απότερες περιφέρειες, τα, τις νήσους, Έχουμε την ανακοίνωση εκείνη για τον θαλάσσιο τουρισμό, τον παράκτιο τουρισμό και εκεί έχουμε προσέγγιση με τους κόμβους, κλάστερς, περιφερειακή προσέγγιση. Το Μάρτιν, αν δεν κάνω λάθος, θα αρχίσει ένας πανευρωπαϊκός διάλογος με τις λιμενικές αρχές σε όλη την Ευρώπη. Ατλαντικό, Βαλτική, νησιά, ξέχασα να το πω υπάρχει αυτή η ανακοίνωση. Πέρσι εγκριθήκε. Ευχαριστώ για την υποστήριξή σας. Είμαι στη διάθεσή σας για συνάντηση με Task Force, Intergroup, ό,τι θέλετε. Θα διαβάσω όσο είπατε στην κυρία Επίτροπο και ελπίζω να τα ξαναπούμε στο άμεσο μέλλον εδώ στην Επιτροπή σας. Σας ευχαριστώ πολύ. και τώρα ο κύριος Αντιπρόεδρος. Νομίζω ότι η τελευταία μισή ώρα έδειξε ότι είναι πάρα πολλά πράγματα τα οποία πρέπει να αντιμετωπίσουμε στον τομέα του τουρισμού. Η ελπίδα μου είναι ότι με συνεργασία και με τον κύριο Ορτούν και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορούμε να προωθήσουμε το θέμα αυτό. Έχουμε λοιπόν μια σημαντική πρωτοβουλία, ένα πρόγραμμα που αναφέρεται ως επιτόπιος τουρισμός, αυτός είναι ο τίτλος του, και η ελπίδα μου είναι ότι θα μπορέσουμε να έχουμε μια καλή συνεργασία με όλους τους ενδιαφερόμενους και τον κύριο Ορτούν τους επόμενους μήνες. Θέλω ε, τέλει να πω ότι είπαμε πολλά για τους Κινέζους τουρίστες. Τις επόμενες εβδομάδες, τους επόμενους μήνες, τους επόμενους ε, χρόνους θα είναι σημαντικό το θέμα του κινέζικου τουρισμού και νομίζω θα είναι χρήσιμο να υποδεχτούμε και μια αντιπροσωπεία που θα έρθει εδώ από Κινέζους επιχειρηματίες. Νομίζω ότι μπορείτε να υποστηρίξετε και αυτή την ε, πρωτοβουλία. Ελπίζω ότι οι συντονιστές θα βρουν τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να εξασφαλίσουμε μια καλύτερη <clears throat> επαφή με τους Κινέζους αυτούς εκπροσώπους. Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ και ο Πρόεδρος. Έχει τελειώσει λοιπόν η πρώτη συνεδρίαση της Task Force για τον τουρισμό. Και μπορούμε να περάσουμε στο τέταρτο σημείο της τη διάταξης και θέλω να χαιρετήσω τον κύριο Ντάνιελ Ντέλτον από την ECR, ε, από το κόμμα το συντηρητικό και μεταρρυθμιστικό στην Επιτροπή μας. Καλώς ήρθατε. Εντάξει. Παίρναμε λοιπόν στο επόμενο σημείο, το σημείο 4, βάρος και μέγεθος <clears throat> των ε, οχημάτων για διεθνείς μεταφορές και δίνω αμέσως το λόγο στον κύριο Λάιχτφριντ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ένα λεπτό να αποχωρήσουμε όσοι θέλουν λέει ο Πρόεδρος. Ich glaube, jetzt kannst ξεκινήσετε. Α, σας κατευχαριστώ. Συνάδελφοι, ευχαριστώ. Καταρχήν για τη μεγάλη στήριξη στις διαπραγματεύσεις αυτές με το Συμβούλιο και την Επιτροπή που δεν ήταν εύκολες. Ήταν αντίθετα πολύ λεπτό το θέμα, αλλά τελικά πετύχαμε και από ό,τι κατάλαβα ήταν εκεί και όλοι οι σκιώδεις και θα σας πω το αποτέλεσμα. Ασχοληθήκαμε με διάφορα θέματα, τα καλά νέα είναι ότι το διαμεθοριακό θέμα ήταν ίσως το σπουδαιότερο και αποφασίσαμε όπως είχε αποφασίσει και το Κοινοβούλιο, ταυτίστηκε σχεδόν με τη θέση μας και το Συμβούλιο, επομένως είναι σαφή τα πράγματα. Όποτε χρησιμοποιούνται μεγαλύτερα, βαρύτερα, ψηλότερα, μακρύτερα φορητά, μπορεί να υπάρξουν προβλήματα, αυτό ισχύει όμως για όλη την Ευρώπη, όχι μόνο για τη Βόρεια. Το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ισλανδία είναι κάπως ιδιαίτερο το πρόβλημα και γύρω από αυτό επικεντρώθηκαν τα υπόλοιπα. Θα σας τα πω σημείο σημείο για να τα καταλάβετε καλύτερα. Στο θέμα πιο βιώσιμων μοτέρ κινητήρων Κομισιόν δέχτηκε την πρότασή μας για τη χρησιμοποίηση και εναλλακτικών καυσίμων και εμείς δεχτήκαμε ότι για τα βιοκαύσιμα και τα συνθετικά καύσιμα δεν χρειάζεται να γίνει τίποτα ιδιαίτερο. Επίσης συμφωνήσαμε για τα λεωφορεία σε πολλά τμήματα. Μέχρι τώρα η κυκλοφορία κοντέινερ 45 ποδών ήταν πολύ δύσκολη, τώρα διευκολύνθηκε. Θα μπορούν να έχουν 15 παραπάνω εκατοστά τα φορτηγά, οι πλατφόρμες τους για να αποχωρούν και αυτά τα containers. Και τέλος θεωρήσαμε λογικό να μπορούν να χρησιμοποιούν και αυτά και μικρότερα κοντέινερ. Αλλιώς οι μεταφορείς αγαθών θα έπρεπε να αγοράζουν για κάθε τύπο κοντέινερ χωριστές πλατφόρμες φορτηγών. Επίσης, ήταν, θεωρήσαμε ενδιαφέρον το εξή. Ζητήσαμε από την Κομισιόν να κάνει αναθεώρηση του όλου ορισμού των συνδυασμένων μεταφορών και από τις πιο ενδιαφέρουσες συζητήσεις ήταν το θέμα της αεροδυναμικής όπου χωρίστηκε η συζήτηση σε δύο τμήματα, τα μπροστινά και τα πισινά. Συμφωνήσαμε για το μέγιστο μήκος των αεροδυναμικών τμήματων σε 200 χιλιοστά. Γιατί έτσι μπορούν να ανεβούν τα φορτηγά και στους σιδηροδρόμους και από την άλλη συμφωνήσαμε έναν πολύ πολύπλοκο κατάλογο κριτηρίων που ήταν ουσιώδης για μας και δεχτήκαμε να μην γίνει με κατεξουσιοδότηση πράξης αλλά δεν έχει αυτό κανένα πολιτικό, καμία πολιτική επίπτωση ή κόστος. Η δυσκολότερη συζήτηση που σχεδόν απέτυχε, κόντεψε να αποτύχει, ήταν το θέμα του αεροδυναμικού καλύματος. Mm. Το ήθελαν υποχρεωτικό και η λύση που βρέθηκε ήταν συμβιβασμός δηλαδή. Να είναι δυνατόν να εφαρμόζονται αυτά τα καλήματα μόλις υπάρξουν Αλλά για να γίνει αυτό χρειάζεται πρόσθετη νομοθεσία και αυτό ήταν το πρόβλημα από την αρχή. δηλαδή ο τύπος έγκρισης που πρέπει να αλλάξει ώστε να μπορούν να μπουν αυτά τα καλύματα. Και κάτι σημαντικό πανευρωπαϊκό είναι ότι αν μια χώρα μέλος θέλει να αλλάξει κάτι δεν έχει πρόβλημα. Αλλά το θέμα είναι η πανενοσιακή αλλαγή. Και ο συμβιβασμός ήταν ότι πρέπει να εφαρμοστεί αυτή η αλλαγή τρία χρόνια μετά από μεταβατική περίοδο τριών ετών και υπάρχει υπόσχεση της Κομισιόν να κάνει αυτή την πρόταση μετά από τρία χρόνια. Αυτό έχει δύο πλέον εκτήματα. Επιταχύνεται η νομοθετική διαδικασία που πρέπει να εφαρμοστεί αλλιώς δεν ξέραμε πότε θα έκανε την πρότασή της και έπειτα να είναι γρήγορη αυτή η εφαρμογή των καλύπτρων γιατί πολλές εταιρείες κατασκευής φορτηγών δεν τα θέλαν αυτά τα κάλυπτρα. Δική μας επιτυχία ήταν όχι δική τους θα έλεγα και απ' την άλλη αν πολλές χώρες μέλη θέλανε νωρίτερα να εφαρμόσουν τα αεροδυναμικά αυτά μέτρα που είναι ιδιαίτερα σημαντικό θέμα στο Ηνωμένο Βασίλειο και σε μεγάλες πόλεις όπως το Λονδίνο λύθηκε και αυτό. Για το θέμα των συγχυσμάτων πάνω στα φορτηγά θα μπορούν τα κράτη-μέλη να επιλέγουν όποιο σύστημα θέλουν. Αλλά τελικά αν έχει ζυγαριά το φορτηγό τότε πρέπει η ζυγαριά αυτή να μπορεί να επικοινωνεί με τον οδηγό Ε, ακούγεται εύκολο αλλά είδαμε ότι όλα τα νέα φορτηγά έχουν κάποιο είδους ζυγάρια στο λεγόμενο keybox τους που δεν το καταλαβαίνω ούτε εγώ λέει ο μιλητής για να γνωρίζει το φορτηγό κάθε φορά πόσο φορτίο έχει και να παρέχει την πληροφορία αυτή στον οδηγό. Αυτό θέλαμε. Τα νέα φορτηγά να έχουν αυτές τις ζυγαριές που να πληροφορούν τον οδηγό. Τέλος, καταφέραμε αυτό που ήθελε το Κοινοβούλιο, την ρήτρα αναθεώρησης, τρία χρόνια μετά την εφαρμογή και με της οδηγίας. Αυτά. Η περίοδος μεταφοράς είναι 24 μήνες τις οδικές και από το 17 θα αρχίσουν να ισχύουν όλα αυτά και τελικά δύο χρόνια κράτησε η διαπραγμάτευση μου φάνηκαν πέντε αλλά ήταν δύο και νομίζω ότι τώρα πάει. Τελείωσε. Congratulations. And now Wim van... Ε, συγχαρητήρια Σας ευχαριστώ, λέει και ο Βλέπω από τον κύριο Λάιχτφριντ πόσο δύσκολο ήταν το θέμα γιατί γκρίζεραν και τα μαλλιά του. Δύο χρόνια εργάζεται για το θέμα αυτό ως εισηγητής δύο χρόνια που τον έκανα να γεράσει πέντε χρόνια. Κύριε Λάιφτριτ, για τα αποτελέσματα της εργασίας αυτής. Εγώ είμαι συντονιστής από το ΕΛΚ, αλλά είμαι και Ολλανδός και οι Ολλανδοί τη βρίσκουν με τα μεγάλα καμιόνια. Δεν είναι κάτι το οποίο ακριβώς αυτό που θέλαμε, αλλά νομίζω ότι είναι μια καλή κίνηση. Τώρα υπάρχει μια κάποια σύγχυση σε ό,τι αφορά αυτό το σχέδιο σύστασης. Σας λένε ορισμένοι και ο κύριος Λάιχτη τροποποίησε το κείμενό του σε σχέση με αυτά που ελέγχθησαν, αλλά νομίζω ότι αυτά τα οποία βρίσκονται τώρα στο, στο κείμενό του είναι συμβιβαστικές λύσεις οι οποίες έχουν προέλθει από τον τριγωνικό διάλογο δεν θα πρέπει να νομίζετε ότι αυτά είναι οι προτάσεις του κυρίου Λάχφρυντ Είναι το κείμενο συμβιβασμού στο τριγωνικό διάλογο. Έτσι κατάλαβα. Αν είναι διαφορετικά, πέστε μου το. Εγώ πιστεύω ο Ισμαήλ να μου μεταφέρει ένα πιο εύκολο φάκελο. Ευχαριστώ λέει ο Ισμαήλ Ερτού. Και από τη δική μου πλευρά τώρα Μα πρώτα τους κύριους συγκητές να ακούσουμε και μετά τον κύριο Ερτού. Σας ευχαριστώ. Και από τη δική μου πλευρά θέλω να συγχαρώ τον κύριο Λάιχτ Φρίντ για το χρόνο και την προσπάθεια που έχει δαπανίσει για το θέμα αυτό. Είναι ένα πολύ δύσκολο ζήτημα. Ξεκίνησε λοιπόν με το θέμα των, ε, <clears throat> των οικοκόμπι όπως λένε. Αυτό είναι μια έννοια που στις κάτω χώρες ε, έχει ισχύει εδώ και 20 χρόνια τουλάχιστον. Είναι καλό για το περιβάλλον, είναι καλό και για, το, για την οικονομία καυσίμων. Έχει μειώσει τη χρήση έχει μειώσει τον αριθμό των ατυχημάτων η έννοια των οικοκόμπης, αλλά επειδή ξεκίνησε με τα θέματα αυτά θα ήθελα να ξέρω ακριβώς ποια είναι η άποψή του για το θέμα αυτό. Ίσως χρειάζεται να του μιλήσω προσωπικά. Το ξαναλέω, θα ήθελα να μας πει ο κύριος ε, ο κύριος και, η, και η γραμματεία ποια είναι η τελική θέση στην οποία καταλήξαμε για τα μεγάλα αυτά τα φορτηγά, τα eco combis. Το παράτημα 2. Στο παράτημα αυτό ο κύριος ε, Λάιφτριτ έχει μεταφέρει τις προϋποθέσεις για τα μεγάλα αυτά φορτηγά, τα μακριά φορτηγά, τα εκοκόμπης, τα οποία προέρχονται από το κείμενο του Συμβουλίου. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν αυτό το θέμα των γιγαντίων φορτηγών των εκοκόμπης. Υπάρχουν όμως προβλήματα που αυτά τα φορτηγά, παραγωγή χάρη αυτά τα οποία μεταφέρουν δρεπτά άνθη, δεν μπορούν να μπουν στη Γερμανία γιατί <clears throat> απαγορεύεται η κυκλοφορία τους λόγω περιβάλλοντος. Θα ήθελα λοιπόν να ξέρω τι ακριβώς προβλέπει το κείμενο του κυρίου Λάιτφριτ για το παράδειγμα 2, για τα μεγάλα αυτά φορτηγά, τα εκοκόμπης. Θα ήθελα λοιπόν να ακούσω και από τη Γραμματεία ποια ακριβώ ήταν η θέση του Συμβουλίου σε αυτό το τριγωνικό διάλογο. Ο κύριο Λάιφρυντ θα έχει το λόγο στο τέλο, έτσι κι αλλιώ, λέει ο πρόεδρο. Η Γκεζίνε Μάισνερ, σα ευχαριστώ κύριε πρόεδρε. Και από τη δική μου πλευρά θα πρέπει να εκφράσω τι ευχαριστίε μου στον κύριο Λάιφρυντ, ο οποίο ω εισηγητή έκανε πάρα πολύ σημαντική εργασία. Ξέρουμε ότι έκανε πολλή προσπάθεια και καταλήξαμε και στον τριγωνικό διάλογο σε ένα αρκετά σημαντικό συμβιβασμό για τα μεγάλα αυτά φορτηγά και τόνισε ο κύριος Λάχρυντ ότι εκεί που υπάρχουν κανόνες σε ορισμένα ευρωπαϊκά κράτη θα πρέπει να διατηρηθούν. Αυτά μπορείτε να δείτε και στο διαδίκτυο. Εμείς προσπαθήσαμε να βρούμε μια λύση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και υπάρχει και το θέμα της καμπίνας του οδηγού για τα φορτηγά αυτά. Πρέπει να υπάρξει και μια ευρωπαϊκή λύση η οποία να ισχύει σε όλη την Ευρώπη. Θα πρέπει να βρούμε και εδώ μια λογική λύση και να ισχύουν οι ίδιοι κανόνες. Τώρα το θέμα του, των παρελκομένων ήταν κάτι στο οποίο δεν υπήρξε καμία συμφωνία. Νομίζω ότι γενικά μου η συμβαστική λύση η οποία, στην οποία καταλήξαμε είναι θετική και μπορούμε εκεί να ε, θα πρέπει να κάνουμε και μια να ακούσουμε και από την Κομισιόν να μας δώσει η Κομισιόν μια έκθεση για αυτά τα μεγαλύτερα φορτηγά γιατί αυτό απαιτεί και μια διαβούλευση από όλους αυτούς οι οποίοι εργάζονται στον τομέα των μεταφορών με φορτηγά αυτοκίνητα και θα ήταν πολύ σωστό να υπάρξει μια τέτοια έκθεση που περιλαμβάνει τι απόψει όλων. Και νομίζω ότι παρά το γεγονό δεν πετύχαμε όλα αυτά που θέλουμε, ήταν πολύ θετικά. Μα έτσι γίνεται στου ε, τριλόγου, λέει και ο πρόεδρο τη Μαρία ε, λέουν Σα ευχαριστώ, αγαπητοί συνάδελφοι. Ευχαριστώ πολύ κύριε Λάκφριντ. Πάρα πολύ χρήσιμα τα όσα κάνατε. Νομίζω ότι έτσι μπορεί να επιληθεί το πρόβλημα όσον αφορά τις διαστάσεις, όσον αφορά το βάρος. Ε, τα κάνατε όλα αυτά με μεγάλη, μεγάλο ενδιαφέρον, μεγάλη όρεξη και επομένως θα πρέπει να λέμε υπόψη τι γίνεται με την υπόθεση της επιμελητίας, τα logistics, τι γίνεται με την μεταφορά. Αυτό είναι κάτι που αφορά όλους τους Ευρωπαίους. Ναι, κάθε ευρωπαϊκή χώρα ε, έχει άλλες ανάγκες, οπότε χρειάζεται οι μεταφορές να μπορούν να προσαρμοστούν σε αυτές τις διαφορές. Στη δική μας χώρα και εμείς έχουμε να διανύσουμε μεγάλες αποστάσεις. Δεν μπορούμε να έχουμε σιδηρόδρομο παντού. Ή καμιά φορά δεν, δεν γίνεται, δεν είναι εφικτό ή δεν είναι συμφέρον οικονομικά. Άρα χρειάζεται κάποια προσέγγιση ε, ευέλικτη. Να έχουμε τη δυνατότητα να μεταφέρουμε περισσότερα εμπορεύματα, αλλά ταυτόχρονα το κάνουμε με τρόπο που να μην βλάπτει το περιβάλλον. Δεν μπορούμε να αναγκάσουμε τις χώρες να έχουν την ίδια προσέγγιση αλλά ελπίζω ότι στο μέλλον θα γίνει αποδεκτό το ότι υπάρχει διαφορετικότητα. Από την άλλη μεριά και η ανταγωνιστικότητα είναι διαφορετική σε κάθε μέρος. Ας βρούμε μια κοινή λύση, ας βρούμε ένα κοινό μοντέλο. Δεν μπορώ παρά να ευχαριστήσω όλους όσους συνεργάστηκαν για αυτή την προσέγγιση που ήταν τόσο επαγγελματική. Είναι μια πρόκληση να είμαστε ανταγωνιστικοί στην επιμελητία. Είναι θέμα πραγματικό. Θα πρέπει να βρούμε μια κοινή απάντηση. Δεν είναι δυνατόν, όπως είπαμε, για το καπάκι εκείνο, δεν είναι δυνατόν να έχουμε ένα καπάκι για όλα, ούτε να έχουμε ένα καπέλο για όλους. Και, και εγώ αν είναι ακόμα το καπέλο, πάλι δεν είναι το να το έχουν όλοι. Εγώ συμφωνώ λοιπόν κάτω από τις προϋποθέσεις αυτές που αναφέρεται και η Στέλλα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ε, ο Evans. Ευχαριστούμε τον κύριο Λάιχτφριντ για τις εξαιρετικές του προσπάθειες. Πάντως, ε, καμιά φορά είναι, είναι εγωιτευτικό να έχει κανείς ε, γκρίζα μαλλιά. Πάντως ε, οι πράσινοι θα επιψηφίσουν αυτό το κείμενο κατόπιν του τριλόγου. Δεν θα κάνουμε τροπολογίε, πάντω σας επαναλαμβάνω ότι για τη δική μας ε, πολιτική ομάδα το θέμα το διασυνοριακό είναι το πιο κρίσιμο. Νομίζω επομένω ότι θα πρέπει να ξεκαθαριστούν κάποια ζητήματα. Τώρα. Θα δούμε πώς θα έχει ο σχεδιασμός το design των ταξί. ή, ή της καμπίνας εκεί όπου είναι ο οδηγό του φορτηγού. Και εκεί θα πρέπει να σας πούμε τις προτάσεις μας. Ευχαριστούμε ο Πρόεδρος. Έχει το λόγο κύριε Άντερσον. Νομίζω ότι έχει σημειωθεί πολύ σημαντική πρόοδο και ευχαριστούμε πάρα πολύ τον ε, εισηγητή αλλά και όλου όσου συνεργάστηκαν μαζί του. Πάντω ευχαριστούμε τον εισηγητή για τα όσα είπε για το Λονδίνο και το ότι χρειάζεται να προχωρήσουμε. Και όσον αφορά το τα ασφαλέστερα φορτηγά, ε, τότε, τότε πρέπει να δούμε τι γίνεται και με την κινητικότητα στι πόλει και για πόλεις, όχι μόνο για, σαν το Λονδίνο, για πάρα πολλέ πόλει στην Ευρώπη. Πάντω ε, στο Λονδίνο ειδικά Έχουμε πολλά πρέπει να βελτιωθούμε όσον αφορά τα φορτηγά. Παρά το ότι έχουμε κάνει πολλά. Ε, είδατε τι με αυτό το μέσο όρο των τριών ετών, γενικά όσον αφορά την ασφάλεια, έχουμε 980 πεζούς οι οποίοι σκοτώθηκαν ή στραφτήκαν σοβαρά. Μέσο όρο στο Λονδίνο τελευταία τριετία. Και 577 ποδηλάτε. μέσο όρο ετησίω. Νεκροί και βαρέω τραυματίε. και οι περισσότεροι τραυματισμοί προκαλούνται από φορτηγά και τραυματισμοί και θάνατοι. Άρα έχουμε ακόμα πολύ δρόμο μπροστά μας ώστε να έχουμε ασφαλή φορτηγά στις πόλεις. Και επομένως πρέπει να δράσουμε από κοινό. Άλλωστε έχουμε και δημοτικές εκλογές την επόμενη διετία στο Λονδίνο. Άρα θα πρέπει αυτό το θέμα να μπαίνει συνεχώς προς συζήτηση και ξέρω πρόβλημα πολλών ε, πόλεων στη κοινό πρόβλημα. Ε, σε κάποιες πόλεις, αλλά όχι παντού, έχουμε περιορισμούς, έχουμε ειδικέ λωρίδες για τα φορτηγά, ε, ειδικέ ώρες για τα φορτηγά. Τέλο πάντων θα πρέπει στις πόλεις κανείς να κοιτάει όλες τις λύσεις, να αξισορροπεί το, τη λύση με τα οικονομικά θέματα που υπάρχουν, τελικά να είναι πιο ασφαλής η πόλη για πεζούς και για ποδηλάτες. Φώστερ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρο και πάρα πολλά ευχαριστώ στο Γιώργο Λάιντφριντ. Ήταν δύσκολο το θέμα αυτό και νομίζω ότι το έργο το οποίο έχει γίνει στον τριγωνικό διάλογο και μεταξύ των Υπουργών Μεταφορών μαζί με τον εισηγητή ήταν πάρα πολύ σημαντικό και φυσικά είναι και σημαντική η υποστήριξη των σχεδόν εισηγητών. Είναι πολύ καλό το αποτέλεσμα. Φυσικά πολλά από αυτά τα θέματα είναι συναισθηματικού χαρακτήρα φορτισμένα και κρατούν πάρα πολύ χρόνο και για, την, ε, ε, το σχεδιασμό της καμπίνας οδηγού θα πρέπει να, να οδηγηθούμε σε μια νομοθεσία που οδηγεί σε έγκριση τύπου. Νομίζω όμω ότι με την προσπάθεια του κύριου Λάιφρυντ έχει ασκηθεί πίεση και στους κατασκευαστές φορτηγών και νομίζω ότι ήταν ένα πολύ καλό αποτέλεσμα της προσπάθειάς του. Χαίρομαι λοιπόν ότι κατέστη δυνατόν να ρυθμιστεί και το θέμα του Ηνωμένου Βασιλείου, δεν ήταν θέμα για τα άλλα κράτη-μέλη. Για μας όμως ήταν πολύ σημαντικό. Θέλω να ευχαριστήσω τον εισηγητή που επέλυσε το θέμα αυτό και τέλος για τα ζητήματα επικορικότητας. Αυτό ήταν πάντα εμπλεκόμενο στο ζήτημα αυτό και φυσικά αυτό ενδιαφέρει τους Ιρλανδούς, αλλά τα διαμεθοριακά προβλήματα ήταν το πώς θα μπορέσουμε να έχουμε μια συμφωνία. Αν υπάρχει ένα φορτηγό 60 τόνων θα πρέπει να έχει έγκριση και πέραν των εθνικών συνόρων. Από τη δική μας ε, πλευρά λοιπόν, από την Βρετανική πλευρά που έχουμε ένα νησί με μεγάλη κίνηση φορτηγών, δεν θέλουμε τα μεγάλα φορτηγά. Καταλαβαίνω ότι έχει νόημα για χώρε όπω η Σουηδία και η Φιλανδία, αλλά δεν το θέλουμε εμεί. Έχετε κάνει λοιπόν πολύ καλή εργασία, κύριε Σιγητά, και σα ευχαριστώ και εμεί σίγουρα θα σα υποστηρίξουμε ω ECR και Βρετανική Συντηρητική ε, Αντιπροσωπεία και ο κύριο Φαντάλεν έκανε ορισμένε ε, ε, ερωτήσει προ εσά, αλλά εμεί είμαστε πολύ ικανοποιημένοι. Ο Ισμαήλ Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και από τη δική μου πλευρά θέλω να ευχαριστήσω τον εισηγητή ο οποίος διέλαβε ένα πάρα πολύ δύσκολο ζήτημα και ήταν φανερό από την αρχή το αποτέλεσμα το οποίο έχει επιτευχθεί κατά τη δική μου άποψη είναι απόλυτα αποδεκτό Μα φυσικά έπαιξε μεγάλο ρόλο η για να φτάσουμε στο σημείο αυτό. Και τώρα αν πρέπει να νερώσω λιγάκι το κρασί αυτών που είπαν ορισμένοι άλλοι, τα πράγματα θα είχαν πάει πολύ καλύτερα αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν προσπαθούσε με το ζόρι να επιβάλλει αυτά τα μεγάλα φορτηγά. Το γεγονός είναι ότι τα διάφορα θέματα, η καμπίνα του οδηγού, τα ζητήματα των αεροδυναμικών εξαρτημάτων μπόρεσαμε να τα αντιμετωπίσουμε σωστά. Η ρύθμιση για να υπάρχει ε, το παράδειγμα της ουράς που φτάνει μέχρι 50 εκατοστά ήταν πολύ θετικό επίσης και με τον τρόπο αυτό έχουμε μια προσθέμενη αξία που από τη δική μας πλευρά δεν είναι ίσως η βέλτιστη αλλά ως συμβαστική λύση είναι πολύ σημαντική. Υπάρχει και μια ρήτρα αναθεώρησης. Ελπίζουμε ότι θα μπορέσει να γίνει το ταχύτερο δυνατόν μια <clears throat> αναθεώρηση. Τρία χρόνια είναι πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα μέχρι να ξεκινήσει η διαδικασία έγκριση τύπου. Θα ήθελα τώρα να αναφερθώ σε ένα άλλο σημείο για τις διαμεθοριακές ε, μεταφορές. Δεν ξέρω αν διαφωνούμε με τον κύριο Φαντάλεν ή όχι, αλλά νομίζω ότι έχει δίκιο ότι πράγματι για τις μεταφορές που περνούν τα σύνορα δεν θα είναι εφικτές όταν μια χώρα επιτρέπει τα μεγάλα φορτηγά και η γειτονική χώρα αν δεν το επιτρέπει καταλαβαίνω ότι σε αυτήν την περίπτωση δεν μπορούν να κινηθούν τα φορτηγά. Αυτό έχει να κάνει και με τη Γερμανία. Αυτό είναι ένα θέμα που δεν το έχει διαλευκάνει όπως συνήθως η Κομισιόν θα ήθελα να καταλάβω τι γίνεται από την πλευρά της Κομισιόν. Στην Γερμανία γίνονται έρευνες επιτοπίως για τα θέματα αυτά και αυτές οι μελέτες θα πρέπει κάποια στιγμή να περατωθούν. Αλλά γίνεται συνέχεια μία παράταση αυτών των ε, μελετών και των ε, πειραμάτων. Μα με τον τρόπο αυτό δεν λύνει. το πρόβλημα, απλώς το παρατείνουμε. Θα πρέπει να υπάρξει λοιπόν μια σαφής ερμηνεία της νομοθεσίας. Θα πρέπει όμως να καταλάβουμε τι ισχύει για διαμεθοριακές μεταφορές και θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι στις ε, πυκνοκατοικημένες περιοχές να μην υπάρξουν προβλήματα και αν μπορούμε να αφήσουμε τις πόλεις απ' έξω και να αντιμετωπίσουμε μονάχα τη μετακίνηση στου αυτοκινητοδρόμου, αυτό θα είναι θετικό. Και ούτως ή άλλως νομίζω ότι ο εισηγητής επέτυχε ό,τι μπορούσε ανθρωπίνως να επιτευχθεί. Η Ίνες Αιάλα ο εισηγητή Ευχαριστώ. Και ανθρωπίνω να επιτευχθει η Ινε Αγιάλα σεντερ ευχαριστω και εγω να συγχαρω τον εισηγητή. Ήταν δύσκολη δουλειά, κράτησε πολύ χρόνο. Ε, ήδη υπήρχε ένα status quo και το πρόβλημα ήταν ότι ήθελε η Επιτροπή να ανατρέψει αυτό το status quo, οπότε έπρεπε να έχουμε καινούριου ε, νόμου, καινούριου κανόνε που βρήκαν άλλου σύμφωνου και άλλου όχι. Τι να σας πω, με σοκάρισε κάπως ε, αυτό που ε, πρότεινε ο εισηγητής στην οδηγία με το όνομά του. Δεν καταλαβαίνω. Τι εννοεί. φανταστείτε ο καθένας να ονομάζει την οδηγία για την οποία είναι εισηγητής με το όνομά του. Τι να πω εγώ, που έχω να... Και τι θα γίνει, εγώ έχουμε κάτι για τα πρόστιμα, θα, θα μας πάρουμε τις πέτρες. Πάντως κατεβλήθη σημαντική προσπάθεια. Είχαμε καθυστέρηση, αλλά τελικά έχουμε τώρα κάποιο είδου προσπάθεια προσαρμογής και με αυτό το πλέγμα διατάξεων να δούμε πώς θα αλλάξει η δυναμική της κατάστασης των φορτηγών να έχουμε κάποιες καμπίνες ασφαλέστερες. Ασφαλέστερες και για τους φορτηγατζίδες αλλά και για τους άλλους χρήστες του δρόμου. Και έτσι σε περίπτωση ατυχήματος να είναι τα πράγματα καλύτερα για τους πεζούς. Έστω και με καθυστέρηση επομένω, έχουμε αυτή την πρόταση και έχουμε κάποιες τεχνικές αλλαγές όπως και στην ασφάλεια των καμπίνων για τους ευάλωτους πεζούς. Αυτό όμως δεν είναι μόνο τεχνικό θέμα. Είναι κάτι παραπάνω. Επίσης να σας πω ότι θα ήθελα κάπως απλά να μου εξηγηθεί τι γίνεται όσον αφορά το πέρασμα των συνόρων. Θα είναι ευκολότερα τώρα τα πράγματα. Να μην δημιουργήσουμε τώρα με το καινούριο πλέγμα διατάξεων εκείνους τους ε, φορτηγατζίδες οι οποίοι έρχονται από την περιφέρεια της Ένωσης και έχουν δυσκολία στην διάβαση των συνόρων. Ευχαριστώ κύριος ε, Λάιφρυ Α, μια στιγμή. ο εκπρόσωπος της DigiMove. Σε ευχαριστώ πρόεδρε. Θα θέλαμε καταρχήν να υποστηρίξουμε πλήρως το αποτέλεσμα του τριμερούς διαλόγου. Ας μην τα πω ένα-ένα τα καινούργια στοιχεία αλλά μόνο τις νέες τροποποιήσεις για τα φορτηγά ώστε να γίνουν πιο αεροδυναμικά τις νέες συσκευές και για να βελτιωθεί η οδική ασφάλεια. Επίσης θέλω να αναφέρω τις εξαιρέσεις για ορισμένα οχήματα που χρησιμοποιούν ελακτικά καύσιμα και που ναι. επίσης νομίζουμε ότι θα είναι πρασινότερα οχήματα. Ναι. Λυπούμαστε γιατί μερικές πτυχές της αρχικής πρότασης δεν ετέθησαν σε αυτή την αναθεώρηση όπως τους κανόνες που προτείναμε για τη βελτίωση της εφαρμογής για το overload, για την υπερφόρτωση που μπορεί να έχει επιπτώσει στην οδική ασφάλεια αλλά και στην ποιότητα των υποδομών. Θα θέλαμε αυστηρότερους κανόνες, αλλά όπως είπε και ο εισηγητής, το κείμενο είναι αποτέλεσμα συμβιβασμού. Επαναλαμβάνω την πλήρη στήριξη της Κομισιόν για το τελικό κείμενο που έχετε μπροστά σας. Δεν τελείωσε η υπόθεση. Πρέπει ακόμη να συνεχιστούν ορισμένες, να ορισμένες τεχνικές λεπτομέρειες όπως το είδος των εγκρίσεων και ή των εγκρίσεων ανατύπω και ο στόχος είναι να καταλήξουμε σε πρόταση το 16 για τον τύπο των εγκρίσεων ή για τους εγκρίσεις ανατύπω και υπολογίζουμε στη στήριξή σας για την έγκριση και αυτού του τμήματος. Τέλος, θα ήθελα να σημειώσω αυτά που είπε ο κύριος Έρτουκ για τους κανόνες για τη διαμεθοριακή χρήση μακρύτερων φορτηγών. Δεν ετέθη σε αυτή την αναθεώρηση και πράγματι οι κανόνες όσοι έχουν αυτή τη στιγμή ίσως να μην είναι και σαφέστατοι. Αυτό θα το δούμε και αυτό αργότερα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε και τώρα πάλι ο συγητής. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ συνάδελφοι. Κύριε Βαντενκάμπ, φυσικά εγώ δεν μιλούσα για το περιεχόμενο. Ε? normal for a member of this committee. The first phase till we decide. Υπήρξαν δύο φάσεις. Στην πρώτη φάση μετά την απόφαση ήμασταν υποχρεωμένοι να δούμε τι απόφαση θα πάρει το Κοινοβούλιο κατά του Συμβουλίου. Και θέλαμε να περάσουν όσο το δυνατόν περισσότερα στοιχεία. Βασιστήκαμε στη θέση του Κοινοβουλίου. Τι έγινε λοιπόν, θελήσαμε να πετύχουμε όσο το δυνατόν περισσότερα με αυτή τη βάση, αυτή τη βάση, τη βάση αυτής της απόφασης. Για μένα ήταν θέμα αρχή αυτό. Δεν είχα πρόβλημα με την ονοματολογία. Άκουσα όμως σήμερα ότι άλλαξαν οι κανόνες και γι' αυτό. Ίσως στο μέλλον να ξανατέθηκα. για το διαμεθοριακό θέμα οι διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο και την Επιτροπή αποφασίσαμε στην πρώτη ανάγνωση αυτά που αποφασίσαμε στην πρώτη ανάγνωση βρίσκονται τώρα στο συμβιβασμό Λύθηκαν όλα τα νομικά προβλήματα. Νομίζω ναι. Αν κανεί έχει αμφιβολίες να το θέσει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Μέχρι τώρα κανείς δεν διαμαρτυρήθηκε όμως από τους ενδιαφερόμενους. Αν θελήσουν μπορούν. Και εγώ φυσικά είμαι υπέρ του συμβιβασμού που δεν μπορεί πια να τροποποιηθεί. Παρακαλώ όσους τον υποστηρίζουν να μην καταθέσουν και άλλες τροπολογίες. Γιατί θα αγκαστώ να θα απορρίψω. Εφόσον θα απορρίψουν το συμβιβασμό. Σας ευχαριστώ λοιπόν για την υποστήριξή σας μέχρι τώρα και νομίζω εσάς ιδιαίτερα κύριε Πρόεδρε που μας αφήσατε να κάνουμε ό,τι θεωρήσαμε ότι έπρεπε. Κύριε Φαντάλεν, σύντομα παρακαλώ όμω. Πάρα πολύ σύντομα κύριε Πρόεδρε. Έθεσε ένα ερώτημα για το παράτημα 2 και δεν πήρα καμιά απάντηση. <clears throat> Είπα ότι θα ήθελα να έχω μία σαφήνεια και σε νομικό επίπεδο για το παράτημα 2. Παρακαλώ να μου δώσετε αυτή την απάντηση. Θα τα πω γερμανικά λέει ο Το ερώτημα το οποίο έχει θέσει ο κύριος Φαντάλεν πρόκειται για τα παρελκόμενα. Αυτό βρίσκεται στο παράτημα. Υπάρχει ένα παράτημα το οποίο περιλαμβάνει τη θέση του Συμβουλίου και ένα που περιλαμβάνει τη θέση του Κοινοβουλίου. Φυσικά είναι διαφορετικές αυτές οι δύο θέσεις, δεν έχουν φτάσει σε κάποιο συμβιβασμό. Αλλά ούτως ή άλλως το θέμα αυτό δεν έχει τεράστιες συνέπειες σε νομικό επίπεδο. Μπορούμε με τον κύριο Φαντάρε να κοιτάξουμε από κοινού το παράδειγμα εάν θέλετε να έχουμε κάποιες διευκρινήσεις. Αλλά νομίζω ότι όλα αυτά δεν πρόκειται να επηρεάσουν την τελική συμφωνία. Ίσως μπορώ να βοηθήσω κι εγώ στην ε, διευκρίνηση. Ξέρουμε ότι το παράτημα μπορεί να προσθεθεί στο, στην, στο τελικό κείμενο, αλλά αυτό το οποίο είναι νομικά δεσμευτικό δεν είναι το παράτημα. Προσθέθηκε λοιπόν αυτό το παράτημα και εγώ θα ήθελα να, να, να προσαρτηθεί και η απάντηση του κυρίου Σιμ Κάλλας στο ερώτημα που είπα εγώ όπου είπε ο Επίτροπος Κάλλας στο παρελθόν ότι κατά την άποψη της Κομισιόν απαγορεύεται η κυκλοφορία των ε, μεγάλων φορτηγών σε, ευρω... έδαφος χωρών που δεν έχουν εγκρίνει. Βέβαια, έχουμε διαφορετικά πράγματα σε σχέση με το, τη νομική ισχύ των παράτημάτων. Το παράτημα είναι παράτημα, αλλά το κείμενο είναι αυτό το οποίο είναι νομισκά δεσμευτικό για το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο και μέχρι τις 4 Φεβρουαρίου μπορείτε ούτως ή άλλως να καταθέσετε τροπολογίες αλλά δεν θέλουμε να θέσουμε σε κίνδυνο αυτήν την ε, συμβιβαστική λύση. Έχετε κάποιο ερώτημα, ο κύριος Σέρτουχ. Συγγνώμη που επανέρχομαι στο θέμα αυτό, αλλά είχα διατυπώσει και εγώ ένα ερώτημα για τις διάφορες μελέτες ε, επιτοπίως που γίνονται που συνέχεια παρατείνονται χρονικά. Θα πρέπει η Κομισιόν να μας πει τι θα γίνει. Ναι, το ξέρω λέει ο πρόεδρος Κράμερ, αλλά δεν είναι κάτι το οποίο πρέπει να αντιμετωπιστεί σε αυτή τη συζήτηση και εγώ νομίζω ότι δεν έχει νόημα να έχουμε πιλωτικά προγράμματα τα οποία είναι, συνεχίζονται στο διηνεκές. Η Κομισιόν λοιπόν έχει ακούσει αυτά που είπαν οι βουλευτές. Θα πρέπει να καταλάβει η Κομισιόν ότι τα πιλωτικά σχέδια πρέπει να έχουν ένα χρονικό περιορισμό. Λοιπόν, τροπολογίες μέχρι τις 4 Φεβρουαρίου στις 12 το μεσημέρι Ευχαριστώ και πάλι τον εισηγητή και όλους τους σκιώδες εισηγητές οι οποίοι παρά τις διαφορετικές θέσεις έχουν καταφέρει να εργαστούν από κοινού για να σφυριλατήσουν μια κοινή θέση της Επιτροπής μας. Αυτό ήταν ένα καλό δίδαγμα και μπορούμε να είμαστε ικανοποιημένοι με το τελικό αποτέλεσμα. Εντάξει, <clears throat> ερχόμαστε τώρα στο επόμενο σημείο της διάταξης. είναι σύσταση προς την Κομισιόν για τις διαπραγματεύσεις TTIP. Έχουμε τη γνωμοδότηση που θα παρουσιάσει ο Βιμ Φαντεμκάμπ. Και του δίνω μέσα το λόγο. Ε, Όλοι, Πρόεδρε, γνωρίζουμε ότι οι διαπραγματεύσεις για εμπόριο και επενδύσεις TTIP με τις ε, ΗΠΑ είναι θέμα περίπλοκο. δεν ξέρουμε ακριβώς πώς είναι τα πράγματα τώρα, πού βρίσκεται ε, η κατάσταση. Ξέρουμε ότι η Ρεμόνας προσπαθεί να προσδώσει κάποια περισσότερη διαφάνεια. Και για την Επιτροπή Μεταφορών θα προσπαθήσω όσο πιο σύντομα γίνεται να συντάξω το κείμενο το οποίο απαιτείται τη γνωμοδότηση γιατί μιλούμε για πολύ σημαντικά συμφέροντα σε Ευρώπη και είπα Ιδίω για τις μεταφορές. Ισχύει τούτο. Έχω την πρόταση μου έτοιμη και ευχαριστώ να ακούσω τη γνώμη των συναδέλφων. Ευχαριστώ κύριο που έχει το λόγο. Σα ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε για τους σοσιαλιστές. Είναι μια μεγάλη χαρά να μιλήσει κανείς για τα θέματα της TTIP Θέλω να πω ότι αυτό είναι κυρίως μια συμφωνία μεταξύ της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών σε εμπορικό επίπεδο. Αλλά υπάρχουν και μερικά θέματα τα οποία συνδέονται με αυτή τη συμφωνία. Όταν όμως πρόκειται για μια συμφωνία η οποία ξεπερνάει τον εμπορικό τομέα και έχει επιπτώσεις για όλη την ε, Ευρώπη, το να έχουμε διεθνή διαιτητικά δικαστήρια τα οποία μπορούν να ακυρώσουν την εθνική νομολογία και να έχουμε ένα διατλαντικό ε, σώμα το οποίο μας ε, υπαγορεύει πώς θα πρέπει να νομοθετούμε όταν υποσκάπτονται τα πρότυπά μας για την οδική ασφάλεια παραδείγματος χάρη όταν η αμερικανική πολιτική ε, για τις μεταφορές θα μεταφερθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα έχουμε όλα αυτά τα στοιχεία των Αμερικανικών φορτηγών παραδείγματος χάρη έχω την εντύπωση ότι στη δική μας πολιτική ομάδα η κρίση για, το, για την TTIP δεν είναι ιδιαίτερα θετική και θα αναγκαστούμε να καταψηφίσουμε την συνθήκη TTIP εάν η Κομισιόν δεν κατανοήσει ποια είναι η θέση μας και αντιμετωπίσει τη διαπραγματεύση με τις ΗΠΑ με διαφορετικό πνεύμα. <clears throat> Ευχαριστώ κυρία Φώστα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τον Φίμ Φαντεκάμπ για τα όσα ξεκάθαρα αλλά και με πληρότητα ε, Βεβαίω και σε πάρα πολλέ επιτροπέ συζητάτε και ελκύει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η υπόθεση του TTIP. Συμφωνούμε με τα όσα ανέπτυξε ο εισηγητή και στο ECR προβληματιζόμαστε για τα θέματα που αφορούν τις ε, μεταφορές. Πολύ σωστά τα λέει εδώ. Και από πλευρά της επιμελητίας μεταφορών θα πρέπει στην Ευρώπη να ωφεληθούμε από το ότι έχουμε ωραία και περισσότερο διμερές εμπόριο. Οφελεί τις επιχειρήσεις, ε, την απασχόληση κλπ. Τώρα, όσον αφορά τα άλλα θέματα μεταφορών, σας καλώ να θυμηθείτε τις διαπραγματεύσεις με τη ΣΥΠΑ για τους ανοιχτούς εθέρες. Μετά από τόσα χρόνια ακόμα έχουμε προβλήματα για τις υπερπτήσεις στην ΣΥΠΑ. Κάποια θέματα δηλαδή χρονίζουν και δεν λύνονται εύκολα. Να, και στο TTIP μπορεί να γίνει το ίδιο. Κάτι άλλο το οποίο είπε ο Βιμ είναι οι θαλάσσιες μεταφορές, όπου ούτε και έχουν δει αναγνώριση σε κάποια θέματα. Τεχνικά θέματα, συντήρηση, αυτά θα πρέπει να επιληθούν αν θέλουν να έχουμε μια σωστή εμπορική συμφωνία. Έχουμε όμως πολύ δρόμο μπροστά μας. Να παρακολουθούμε επίσης το τι γίνεται στις άλλες επιτροπές για άλλα θέματα. Πάντως ξεκίνησαμε με το δεξιά. Φαντάζομαι και άλλοι συναδελφοί έχουν θέματα να επισημάνουν. Η ΣΥΑΡ κύριε Σιγητά είναι μαζί σας. Η είναι Μάιστερ. Και εγώ υποστηρίζω αυτά που είπε ο κ. Φαντεκάμπ. Είναι ιδιαίτερα εξισορροπημένη η γνωμοδότησή του, αλλά θα ήθελα και εγώ να εκφραστώ εν γέννη για την συμφωνία TTIP όπως είπανε και τα, οι άλλοι σκιώδες εισηγητές είναι ένα τεράστιο θέμα, ήταν πάρα πολύ σημαντικό και στην προεκλογική εκστρατεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Εγώ θα ήθελα να υπάρξει μια προσπάθεια να δούμε ορθολογικά αυτά τα οποία είναι στο τραπέζι της διαπράγματευσης και όχι να έχουμε συναισθηματικές και συγκινησιακές αντιμετωπίσεις. Είναι απαραίτητο να υπάρξει μεγαλύτερη δυνατή διαφάνεια και ο Όρι Ρενίδη το έχει τονίσει αυτό, όπως και η Επίτροπος Μάλστρομ, είναι απαραίτητο να γίνει αυτή η προσπάθεια να υπάρχει και μια πιο ε, μεγάλη διαφάνεια για τα θέματα εδώ και από τα κράτη-μέλη. Τα πρότυπά μας είναι τα δικά μας πρότυπα και δεν πρέπει να τεθούν σε συζήτηση. Αλλά σε ό,τι αφορά τώρα τις μεταφορές, μπορούμε να έχουμε μια πρακτική, πραγματιστική αντιμετώπιση όταν εξασφαλίσουμε να υπάρχει λιγότερη <laughs> γραφειοκρατία στην έγκριση των οχημάτων, αυτό θα βελτιώσει και τις εξαγωγές των ε, ευρωπαϊκών οχημάτων προς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα πρέπει να το δούμε αυτό λοιπόν και στην TTIP. Φυσικά όμως θα πρέπει να υπάρξει σωστή διατύπωση αυτής της ε, ρήτρας. Αν έχουμε λοιπόν μια συμφωνία εμπορικού χαρακτήρα θα πρέπει να συμπεριληφθούν όλες οι περιοχές και αυτό σημαίνει και τις μεταφορές. Υπάρχει ένα σημείο στο οποίο αναφέρθηκε ο Βιμ στις Ηνωμένε Πολιτείες υπάρχει μεγαλύτερη ε, ιδιοκτησία κατά κάποιο τρόπο μέσα σε εισαγωγικά από τις ΗΠΑ. Πολιτείες. Εγώ θα ήθελα να εξασφαλίσω με τη συμφωνία αυτή να μην υπάρχουν διαφορετικές ρυθμίσεις. Οι Αμερικανοί έχουν ε, ένα ιδιαίτερα ε, κλειστό χαρακτήρα σε ό,τι αφορά τη δημιουργία υποδομών. Θα έπρεπε να μπορούν και οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις να συμμετέχουν. Αναφέρθηκε και ο νόμος Jones, ο οποίος είναι και μια ενεξελίξη διαδικασία, είναι και μια μεγάλη ευκαιρία για την Ευρώπη να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε σε διμερές επίπεδο τη συζήτηση αυτή και να μπορέσουμε να περάσουμε τις δικές μας ε, προτάσεις. Είναι πολλά λοιπόν τα οποία μπορούν να εξασφαλιστούν αν έχουμε την κατάλληλη ευκαιρία και στον τομέα των μεταφορών. Ο Μπάς Άικ έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε και Ευχαριστώ και τον αγαπητό μου συνάδελφο που γνωμοδότησε. Ως πράσινοι βεβαίως θα υποβάλουμε μερικές τροπολογίες που θα θέτουν τα γενικότερα προβλήματα του TTIP. Διότι αυτοί που λένε ότι εδώ δεν συζητάμε τα ευρωπαϊκά πρότυπα δεν λένε απολύτως αλήθεια. Διότι ακόμα και η Επίτροπος Μάλστρο μιλάει για νομοθετήματα και πρότυπα μεταξύ είπα και ΕΕ δεν υπάρχουν πια φραγμοί τελωνιακοί τουλάχιστον. Δεν μιλάμε για δρασμούς και τελωνία πια. Μιλάμε για τους λεγόμενους μη δασμολογικούς φραγμούς που εμείς το λέμε νομοθεσία ή διευθέτηση. Αυτό είναι, μην γελιέστε, δεν μπορούμε να λέμε από τη μία τα πρότυπά μας είναι αδιαπραγμάτευτα και απ' την άλλη μιλάμε για νομοθεσία και κανονισμός. Αυτό είναι το θέμα τελικά. Να μην γελιόμαστε ότι δεν συζητιέται. Θα καταθέσουμε λοιπόν μερικές σχετικές τροπολογίες και θα απευθυνθούμε και στην Επίτροπο Μάλμστρομ συγκεκριμένα για τις μεταφορές υπάρχει ένα θέμα για τα αυτοκίνητα που δεν έχει ακόμη προσεχθεί αρκετά. Συνήθως λένε για αυτό το θέμα υπάρχουν πολλά τεχνικά θέματα που θα μπορούσαν να λυθούν μέσω του TTIP. Ναι, τι εννοούμε τεχνικά. Αυτό είναι το θέμα. Μπορεί κάποιος να ονόμαζε τεχνικό, κάποιο που άλλος θα το ονόμαζε πολιτικό. Για τα θέματα της οδικής ασφαλείας θα μπορούσε κανείς να πει δεν παίζει ρόλο αν είναι αμερικανικό ή ευρωπαϊκό το αυτοκίνητο, αλλά γενικά ισχύει ότι ο πεζός είναι σε καλύτερη θέση στην Ευρώπη από ό,τι στην Αμερική λόγω και του design του αυτοκινήτου. Ποιος λοιπόν θα αποφασίσει τι είναι τεχνικό και τι είναι πολιτικό. Είναι κάτι που πρέπει να το προσέξουμε πολύ περισσότερο και να μην είμαστε αφελείς. Και εδώ θα καταθέσουμε τροπολογίες. Μετά, συνάδελφοι με μεγάλη εμπειρία στις μεταφορές, θα ήθελα να ξέρω πόσοι γνωρίζουν τις τεχνικές προδιαγραφές των αυτοκινήτων. Κάθε μήνα προστίθενται. Στη Γενέβη, υπό την Ιούνισε, όπου υπάρχει εναρμόνιση των προδιαγραφών κάθε εβδομάδα σχεδόν. Πηγαίνουν εκεί οι τεχνικοί εμπειρογνώμονες, ίσως θα έπρεπε και εμείς να τους επισκεφθούμε ως Επιτροπή Μεταφορών, για να δούμε τι γίνεται. Γιατί δεν μπορεί ξαφνικά διμερώς το TTIP να τα λύσει όλα αφού τα συζητάει και ο ΙΕ. Από τις 10 μέχρι τις 13 Μαρτίου μπορούμε να πάμε στη Γενέβη γιατί οργανώνεται το Παγκόσμιο Φόρουμ για την εναρμόνιση των προδιαγραφών οχημάτων. Εκεί θα έρθουν και για Ιάπωνες και Κορεάτες. Γιατί λοιπόν να πούμε ότι αυτά θα τα λύσουμε μέσω του TTIP, πράγμα που θα είναι ακόμα λιγότερο διαφανές όταν αγνοούμε ότι υπάρχουν καν τέτοιες διασκέψεις. Σε γνωμοδότηση της Επιτροπής Μεταφορών λοιπόν θα έπρεπε τέτοια θέματα να τα θίξουμε και αυτά είναι θέματα αντικειμενικά άρα μάλλον μπορούμε να συμφωνήσουμε όχι βέβαια με τον συνάδελφο Βοντεκόμπ αλλά με τους άλλους. Ευχαριστώ για τις φιλοπρονήσεις σου στον βήμα ο Αμάτο. Αγιάλα Σέντερ. Ευχαριστώ και εγώ συμμερίζω με τις ανησυχίες που αναφέρθηκαν από τους συναδέλφους. Συγχαίρω τον κύριο Φαντεγκάμπ για τη γνωμοδότηση που μας έχει φέρει. Και νομίζω ότι είναι απαραίτητο να εξασφαλίσουμε κάποια στοιχεία τα οποία θα μας επιτρέψουν να αποφύγουμε τα προβλήματα της ε, διαπραγματεύσης TTIP η οποία καλύπτεται αυτή τη στιγμή από πυκνό πέπλο μυστήριο, κάτι με το οποίο συμφωνούμε. Θέλω όμως να θέσω αυτό το ερώτημα. Η κυρία Μάστρομ μας έχει παρουσιάσει κάποιες θέσεις που έχουν ενδιαφέρον. Θα ήταν χρήσιμο να έχουμε μια συζήτηση μαζί τη. Τονίζω και πάλι ότι για μας είναι πάρα πολύ σημαντικέ οι ρήτρε για το περιβάλλον και οι κοινωνικές ρήτρε, η προστασία των δημοσίων υπηρεσιών όπως βρίσκονται στην Ευρώπη. Φυσικά είναι τελείω διαφορετικό αυτό στην Ευρώπη από τις ΗΠΑ και τα δικαιώματα των ε, επιβατών και επίσης και οι, για την εργασία και προστασία των συνδικάτων. Όλα αυτά λοιπόν είναι πράγματα τα οποία είναι πολύ σημαντικά στην Ευρώπη. Θέλουμε να τις βελτιώσουμε και όχι να τις υποβαθμίσουμε. Και επίσης οι συγκρούσεις μεγάλων επιχειρήσεων είδαμε τις συγκρούσεις μεταξύ Boeing και Airbus στο, τελ, στο παρελθόν. Δεν ξέρω πώς θα μπορέσει να αντιμετωπιστεί αυτό το θέμα, αν υπάρχουν τέτοιες ε, διαμάχες στο μέλλον και φυσικά και το θέμα της ε, ανταλλαγής δεδομένων. Μετά από την επίθεση στο Σαλιεμπτό αυτό ξανά έγινε επίκαιρο, αλλά εκεί υπάρχουν θέματα που όπως είπαμε υπάρχει ο κίνδυνο και για τα εμπορικά στοιχεία που πολλές φορές έχουν πολύ σχέση με τις επιχειρήσεις μεταφορών και στον τομέα αυτό λοιπόν θα πρέπει να υπάρξει μια βελτίωση της, ε, του, κειμένου και να υπάρξουν προϋποθέσεις για να μπορέσει να δοκιμήσει αυτή η διαπραγμάτευση. Μαρία Κίλουν και σας παρακαλώ ζητώ συγγνώμη που δεν της έδωσα το λόγο προηγουμένως. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πρώτα πρώτα. Να ευχαριστήσουμε θερμά τον εισηγητή. Πρέπει να σας υπενθυμίσω κάτι. Αυτό το οποίο πρέπει να γίνει είναι το κείμενο να αντικατοπτρίζει όσο είπαμε προηγουμένω όσον αφορά τη διαφάνεια. Θα πρέπει στο κείμενο να φαίνεται τι καλύπτεται και τι δεν καλύπτεται. Πάντως η Γκουε δεν είναι ενθουσιασμένη όσον αφορά το πώς προχωρούν τα πράγματα στις διαπραγματεύσεις για το TTIP. Ανησυχούμε και δεν μας αρέσει καθόλου η κατάληξη της υπόθεσης όπως διαφαίνεται. Ξέρετε στον κόσμο δεν υπάρχει μόνο το TTIP, γίνονται και άλλα πράγματα. Με και άλλες εξελίξεις, άρα θα πρέπει να έχουμε τα μάτια μας και τα αυτιά μας ανοιχτά γιατί έχουμε μεγάλες αλλαγές. πρέπει να δούμε τι γίνεται τώρα με τις μεταφορές. Θα πρέπει να εξασφαλίσουμε το ότι οι διαπραγματεύσεις αυτές δεν θα υπονομεύσουν το κοινωνικό μοντέλο της Ευρώπης και δεν θα έχουμε κανένα το κοινωνικό dumping. Μιλώ για τον τομέα των μεταφορών. Προσοχή γιατί η εμπειρία μας από παρόμοιες συνδυαματεύσεις με Αμερικανούς είναι πικρή. Μας ανέφερε τα ναυπηγεία ο κ. Φαντεκάμπ. Ξέρετε είχα την ευκαιρία να μιλήσω με τους Αμερικανούς υπευθύνους για τα παγωθραυστικά. Εμείς δεν μπορούμε να τους ε, ανταγωνιστούμε. Και με το Κογκρέσο τελικά δεν μπορούμε να τα βρούμε. Υπάρχει το θέμα της προστασίας του εθνικού know-how, αλλά βέβαια και της προστασίας των εθνικών εργασιακών δικαιωμάτων. Η Κριστίνα έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ τον εισηγητή για τις προτάσεις που έχει διατυπώσει. Είναι εκπληκτικό ότι μπαίνουμε σε διαπραγματεύσεις εμπορικού χαρακτήρα χωρίς όλα τα θέματα που έχουν να κάνουν με τις μεταφορές να έχουν διευκρινιστεί. Κάναμε συζητήσεις με τους διάφορους ε, βιομηχανικούς κύκλους, την αυτοκινητοβιομηχανία, με, την, ε, με τον αεροπορικό κλάδο και υπάρχει το πρόβλημα της πρόσβασης των ευρωπαϊκών ε, επιχειρήσεων στον αμερικανικό χώρο. <clears throat> Όλα αυτά τα θέματα λοιπόν είναι κομβικά για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις για τις απόψεις τώρα που παρουσιάστηκα από τον κύριο Γκλάφιντ για την θέση των σοσιαλιστών. Δεν έχω απολύτω τίποτα να προσθέσω. Προφανώς και εγώ συμμερίζομαι απόλυτα τις ε, ανησυχίες που ανέφερε και όχι μόνο οι σοσιαλιστές βουλευτές έχουν αυτή την άποψη <clears throat> και πέραν αυτών που αναφέρθηκαν Υπάρχει το θέμα των διαιτητικών δικαστηριών που για μας είναι μια μεγάλη πηγή ανησυχιών στην TTIP. Ευχαριστώ. Η κυρία Ανουτού, το εθνικό μέτωπο, φυσικά είναι κάθετα αντίθετο στην συνέχιση των διαπραγματεύσεων για την συμφωνία TTIP. Αν οι <clears throat> διαπραγματεύσει αυτέ προχωρήσουν, αυτό θα είναι ένα κτύπημα εναντίον των οικονομιών και των ελευθεριών μα. Οι Αμερικανοί είναι αυτοί που λένε ότι αυτή η συμφωνία είναι ένα είδο οικονομικού ΝΑΤΟ. Εμεί είμαστε εναντίον λοιπόν τη διεύνηση των συνομιλιών για θέματα μεταφο... στα θέματα μεταφορών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, αντίθετα από τι ΗΠΑ, αρνείται να προστατεύσει αυτόν τον νευραλικό τομέα, ενώ οι ΗΠΑ εφαρμόζουν ε, μεγάλους περιορισμούς σε ό,τι αφορά τη συμμετοχή ξένων κεφαλαίων στις αμερικανικές εταιρείες. Ενώ εδώ γίνεται ακριβώς το αντίθετο. Εμείς δεν έχουμε καμία προστασία για τον τομέα μας. Υπάρχει λοιπόν μια σοβαρή ανισομέρεια μεταξύ των περιορισμών που επιβάλλουν οι Αμερικανοί στις ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρείες και την ελευθερία που έχουν να αλέθουν οι Αμερικανοί στις ευρωπαϊκές εταιρείες. Οι Αμερικάνοι φυσικά θα συνεχίσουν να προστατεύουν αυτόν τον ευραγικό τομέα που είναι η πολιτική του αεροπορία με το να μην δεχτεί να κάνει κάτι τέτοιο η Ευρωπαϊκή Ένωση κινδυνεύει να αυξήσει περισσότερο τα προβλήματα του κλάδου της πολιτικής αεροπορίας στην Ευρώπη που μας στήσεται από την, Κρήτη, την κρίση. Επιτροπή αυτή είναι αρμόδια. Γιατί υπάρχουν θέματα τα οποία είναι στην εντολή μας. Πάντως υπάρχουν και θέματα τα οποία θα μπορούσαν να έχουν φυγεί, αλλά δεν καλύφθηκαν. Πάντως η διευθυντική εντολή δεν αφορά το Κοινοβούλιο, έγινε και διαμορφώθηκε μεταξύ Κομισιόν και, και Συμβουλίου. Εμεί πιστεύουμε στην πρόσκληση προ την Επιτροπή μα πρέπει να έρθει να μα μιλήσει. Αλλά το ίδιο πρέπει να ισχύσει και για του διαπραγματευτέ που κάθε μέρα τα λένε εκεί. Και να δούμε γιατί κάποια πράγματα δεν έχουν καλυφθεί και να μάθουμε πώ συνεχίζονται οι διαπραγματεύσει. Ιδίω όσον αφορά τα πρότυπα σε σχέση πάντα με τα θέματα ενδιαφέροντός μας. Σκεφτείτε, Πρόεδρε, ποιον θα καλέσουμε. Πάντως από ό,τι ξέρω από άλλες επιτροπές, αξίζει να καλέσουμε την Επίτροπο ή και τους διαπραγματεύτες. Οι μεταφορές είναι θέμα που απασχολεί και άλλες επιτροπές, όχι μόνο εμάς. Πάντως, για να λέμε την αλήθεια, δεν θυμάμαι στο πρόσφατο παρελθόν κάποια άλλη συμφωνία, κάποια άλλη τέτοια διαπραγματεύση που να έχει τόση διαφάνεια. Βέβαια, σε αυτό συνέβαλε το Ευρωπαϊκό που πίεσε προς τούτο. Έχουμε ενημέρωση και υλικό από το τι γίνεται εκεί. Τώρα για το σχέδιο γνωμοδότηση νομίζω πάρα πολύ ωραία έχει συνταχθεί. Στις πάντα είχαμε στα θέματα τα δικά μας. Θα μπορούσα να τον βοηθήσω με κάποιες ε, ιδέες, αλλά νομίζω ότι πάρα πολύ ε, καλά τα έχει ισορροπήσει τα πράγματα στο κείμενο και θα πούμε τα υπόλοιπα όταν έρθει εδώ η Επίτροπος. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Λέει κυρία Αντελή, Δεν θα μακρηγορήσω. Αυτό το κείμενο στον αφορά TTIP δεν έχει πάρα πολλά σε σχέση με την πολιτική των μεταφορών. Έτσι κάποια γενικόλαγα μόνο όσον αφορά αερομεταφορές, όσον αφορά θαλάσσιες μεταφορές. Πάντως αυτό που θέλω να σας πω πρώτο είναι ότι κατόπιν των συμφωνιών για τις αερομεταφορές ξέρουμε ότι δεν υπάρχει αμοιβαιότητα. Αυτό είναι κακό. Κακό για τα συμφέροντά μας. Δεύτερον, όσον αφορά τις ιστορικές πλωτές εδώ, Έχουμε κάποια πρόταση όσον αφορά τις ε, επιδόσεις των ε, κινητήρων για το περιβάλλον, των κινητήρων τέλο πάντων μηχανών ε, των, των σκαφών. Προσοχή, γιατί εμεί έχουμε πιο ψηλά στάνταρ του Αμερικανού. Προσοχή, επομένω, κύριε Φαντεκάμπ. Και σα ευχαριστούμε για την εκθεσή σα. Πρόεδρο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την σύστασή του, για τον συντάκτη και θα ήθελα να προσθέσω από την πολιτική μου ομάδα του συντηρητικού ότι όπως και οι υπόλοιποι θεωρώ και εγώ ότι η συμφωνία αυτή με τη ΣΥΠΑ είναι μεγάλη ευκαιρία για τις ευρωπαϊκές μεταφορές, ιδίως σε δύο τομείς αερομεταφορές Πρώτον, όπου δίνεται η δυνατότητα ευρωπαϊκές εταιρείες να απολούν τα εισιτήριά τους εφόσον μία πτήση αρχίζει τελειώνει σε αμερικανική πόλη και έπειτα οι θαλάσσιες μεταφορές όπου προβλέπεται μέχρι τώρα να χρησιμοποιούνται μόνο πλοία που έχουν ιολογηθεί στα Ηνωμένα Πολιτείε και που ανήκουν σε Αμερικανούς ιδιοκτήτες. Σε αυτούς τους δύο τομείς νομίζω ότι μπορούμε να προωθήσουμε περαιτέρω διαπραγματεύσεις ώστε να μην ε, ώστε να υποχωρήσουν οι Αμερικανοί και στην χώρα μου την Πολωνία επίσης πιστεύουμε ότι οι ευρωπαϊκές μεταφορές μπορούν να κερδίσουν πολλά από αυτή τη συμφωνία. Ευχαριστώ. Τώρα, θα ήθελα να τονίσω ότι η συνέλευση των Προέδρων των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών, όπου εκπροσωπώ εγώ την Επιτροπή μας συζήτησε για την TTIP, ο κύριος Βαν ε, έχει δεχτεί τις τροπολογίες που έχω καταθέσει και θέλω να τον ευχαριστήσω και για αυτό το σημείο. Εγώ πιστεύω ότι, ότι υπάρχει πράγματι μια αδικία σε βάρος της Ευρώπης σε ό,τι αφορά την, τις θαλάσσιες και αεροπορικές μεταφορές. Οι, οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν αντιμετωπίζουν την Ευρώπη, Ευρωπαϊκή Ένωση ως οντότητα. Σε όλες τις ε, περιπτώσεις αρνούνται οι Αμερικανοί να δεχτούν την Ευρωπαϊκή Ένωση ως συνομιλτή γιατί έχουν ένα τεράστιο ε, πλεονέκτημα να αφήνουν την Ευρώπη έξω από τέτοιου είδους συμφωνίες. Και έχουμε πει στον πρόεδρο Σούλτς εγώ μπορώ, ξεκινώ να διαπραγματευθώ την TTIP μόνο όταν υπάρξει η αναγνώριση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως θεσμού για τα θέματα θαλασσίων και εναερίων μεταφορών. Είναι απίστευτο να αφήνουμε να έχουν οι Αμερικανοί ένα τέτοιο ε, πλέον έκτημα. Και οι Αμερικανοί δεν έχουν καμία θέληση να αλλάξουν αυτή την κατάσταση. Μπορούμε να είμαστε αισιόδοξοι όσο θέλουμε, αλλά όποιο συζητά με τους Αμερικανούς καταλαβαίνει ότι δεν έχει κανένα λόγο να είναι αισιόδοξο. Δεν πρόκειται λοιπόν μονάχα για, ένα μια εμπορική συμφωνία γιατί έχουμε μεγάλους εμπορικούς φραγμούς. Όλα παίζονται στο επίπεδο της ρύθμισης. Και ξέρουμε περί πρόκειται. Και οι 500.000 θέσεις που ανέφερε ο κύριος Δεγούχτη... ήταν το μόνο όφελος που θα πάρει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα δεν μιλάει κανένας τίποτα για όλα αυτά τα θέματα. Οι Αμερικανοί θεωρούν ότι είναι μια ευκαιρία να κάνουν πολύ καλές δουλειές στην Ευρώπη. Νομίζω δεν θα κερδίσουμε τίποτα. Και πώς έχουν γίνει όλα. Με απόλυτη μυστικότητα. Αυτό είναι απίστευτο. Πρέπει να υπάρχει πραγματική διαφάνεια σε σχέση με τις διαπραγματεύσει. Δεν μπορούμε να πούμε ναι και μετά η Κομισιόν να μας δίνει τα έγγραφα μονάχα κατόπιν εορτής. Είναι πράγματα που έπρεπε να κάνει γίνει ήδη. Και επίσης το θέμα της ε, είναι κράτος δικαίου Πολιτείες και εμείς είμαστε κράτος δικαίου. Δεν χρειαζόμαστε ανεξάρτητα δικαστήρια μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα κανονικά δικαστήρια. Δεν μπορεί να πει μια εταιρεία «Α, έχουν ελάχιστο μισθό οι Γερμανοί και έτσι χάνω λεφτά, οπότε προσφεύγω σε ένα διαιτητικό δικαστήριο». Όχι, είμαστε ένα κράτος δικαίου και ο νόμος πρέπει να είναι να ισχύει για όλους και όχι να αφήσουμε τα κοινοβούλια απ' έξω από το παιχνίδι και να αποφασίζουν κάποιοι άλλοι ούτε μπορούμε να αποφασίζουμε εμεί για όρια εκπομπών και να πούν οι Αμερικανοί όχι αυτό δεν μας βολεύει και να πηγαίνουν σε ένα διαιτητικό δικαστήριο και το ίδιο πράγμα όταν οι Αμερικανοί κάνουν ρυθμίσεις οι οποίες ευνοούν το δική τους βιομηχανία σε βάρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει εδώ να υπάρχουν αποφάσεις σε επίπεδο κοινοβουλίων και όχι ομάδες από ή οτιδήποτε άλλο. <clears throat> Αυτό είναι κάτι λοιπόν το οποίο πρέπει να εξασφαλίσουμε και γι' αυτό εγώ έχω απόλυτο σκεπτικισμό Κυρίως γιατί όπως είπαμε δεν υπάρχουν καθόλου φραγμοί εμπορικοί. Όλα αυτά που εμπλέκονται στη TTIP είναι θέματα ρύθμισης, κοινή ρύθμισης. Δεν πρέπει λοιπόν εμείς να δεχτούμε μια απορρίθμιση σε βάρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν θα πρέπει να δώσουμε στους αντιδημοκράτες να <clears throat> κερδίσουμε αυτό το παιχνίδι. Πάρα πολύ σύντομα η κυρία Μάισνα. Γι' αυτό το λόγο που είπατε ζητώ όταν εσύ βρίσκεσαι στην ε, συνέλευση των Προέδρων των Επιτροπών να τα τονίσεις όλα αυτά τα σημεία. Εάν εσύ τα έχεις αναφέρει όλα αυτά τα πράγματα, δεν θα έπρεπε να, να είχαμε προχωρήσει τόσο πολύ. Εγώ τόνισα ότι ποτέ δεν μου άρεσε αυτή η πρόταση για την TTIP. Εμείς θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε λοιπόν την ευκαιρία στην συνέλευση των Προέδρων των Επιτροπών να αναφέρεις και να αντικατοπτριστεί αυτό το οποίο έχουμε πει μεταξύ μας. Βεβαίως. Είναι σαφές ότι όχι μόνο μεταξύ των επιτροπών αλλά και μεταξύ των πολιτικών ομάδων υπάρχει έλλειψη κοινών ε, θέσεων υποστήριξης. Εγώ είμαι έτοιμος λοιπόν να μεταφέρω την άποψη της, ε, της ομάδας, της ομάδας σας, χωρίς μικρόφωνο μία πρόταση μονάχα. Ναι, με τη διαφάνεια. Μην μας μιλάτε για άκρος απόρριτα κλπ. Αυτά δεν είναι καθόλου αρεαλιστικά. Έχετε όλα τα σχετικά έγγραφα. Δεν ξέρω εάν εκμεταλλευτείτε το ότι σας επιτρέπετε να πάτε στην αίθουσα που υπάρχει όλο αυτό το υλικό. Να καλέσουμε την Κομισιόν. Ακόμα και η συνθήκη προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, ούτε εκεί δεν έχουμε ε, δώσει διαφάνεια σε τίποτα. Δεν είναι ρελίσκο να λέτε τώρα ότι δεν έχουμε διαφάνεια. Όχι. Δεν έχει αλλάξει ακόμα. Υπάρχουν διάφορα επίπεδα μυστικότητας σε ό,τι αφορά την πρόσβαση στα έγγραφα και την αντιγραφή τους. Εγώ προτού μπω σε αυτό το δωμάτιο δεν μπορώ να κρατήσω σημειώσεις, δεν μπορώ να μιλήσω σε κανένα, δεν μπορώ να χρησιμοποιήσω το κινητό μου τηλέφωνο. Αυτό είναι υπερβολική μυστικότητα. Λοιπόν, αυτό πρέπει να αλλάξει. Εγώ θέλω να ξέρω τι γίνεται στα έγγραφα και να έχω τη δυνατότητα να συζητήσω για αυτά. Αν αλλάξουν τα πράγματα, πληροφορήστε με. Και ξαναδίνω και δίνω τώρα το λόγο στην Κομισιόν. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Είμαι επικεφαλής των διαπραγματεύσεων για τις υπηρεσίες, άρα με αφορούν μερικά πράγματα που είπατε, όχι όλα. Δεν θα μιλήσω για όλα τα θέματα που θέσατε εσείς με τις μεταφορές, γιατί ξεπερνάνε τα δικά μου. Θέλω απλώς να πω για ένα θέμα διαφάνειας που τίθεται. Ο, ε, η Επίτροπος Μάλστρομ έχει κάνει μεγάλες προσπάθειες, θα το αναγνωρίζετε κι εσείς, έχει κάνει στις τελευταίες εβδομάδες και μήνες, με την ε, διευθέτηση που υπάρχει για τα reading rooms πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι Η διαπραγμάτευση αυτή είναι πρωτόγνωρη ως διαφάνεια. Ίσως αυτό εννοεί ότι οι άλλες διαπραγματεύσεις δεν είναι, αλλά τέλος πάντων είναι αλήθεια. Και στο τίτυπη για τη διαφάνεια και για την κοινωνία των πολιτών και για τους κοινοβουλευτικούς φυσικά και εθνικός και ενωσιακός είναι πρωτόγνωρο και θα ήθελα να σας πω ότι οι κοινοβουλευτικοί έχουν πρόσβαση σε όλα τα ενωσιακά τονίζω έγγραφα. Θα επανέλθω σε αυτό όταν μιλήσουμε για τις μεταφορές. Ένα από τα θέματα που τέθηκαν στη γνωμοδότηση είναι ότι οι μεταφορές μέχρι τώρα δεν έχουν συζητηθεί. Εγώ διαπραγματεύομαι για τις υπηρεσίες και παρόλα αυτά μπορώ να το μετριάσω αυτό. Όσοι πήγατε στα Reading Room θα έχετε δει ότι ήδη από τον Οκτώβριο του 2013 η Ένωση υπέβαλε δύο έγγραφα στις διαπραγματεύσεις ή δύο non-papers μία για την αερομεταφορές, την άλλη για τις θαλάσσιες, το άλλο για τις θαλάσσιες και αυτά όπως θα δείτε θέτουν πολύ συνοπτικά όχι όλες τις λεπτομέρειες θέματα που θα ήθελε να συζητηθούν η Ένωση το Jones Act, τους ελέγχους στις αερομεταφορές, αλλά και άλλα θέματα, την αεροπορική ασφάλεια κλπ. Θα έλεγα λοιπόν ότι δεν είναι σωστό να λέμε ότι μέχρι τώρα τα θέματα των μεταφορών δεν έχουν παίξει ρόλο στις διαπραγματεύσεις αυτές. Και ισχύει για κάτι που με ξεπερνάει εμένα τις ε, κυβερνητικές προμήθειες. Η πρόσβαση στην Αμερικανική αγορά είπατε ότι είναι ασυμμετρική σε σύγκριση με το δικό μας άνοιγμα. Γιατί όλοι γνωρίζουμε ότι το σύνθημα Buy American είναι πολύ, παίρνεται πολύ σοβαρά υπόψη. Και αυτό αφορά πολλούς τομείς. Όχι μόνο στις υπηρεσίες, αλλά και για τις κυβερνητικές πραμήθειες. Έχουν τεθεί πολλά θέματα μεταφορών και γι' αυτό θεωρώ ότι και αυτό πρέπει να μετριαστεί για να ανταποκρίνεται περισσότερο στην πραγματικότητα αυτά που είπατε. σε σύγκριση και με το ψήφισμα του Μαΐου του 13 του Κοινοβουλίου όπου θέματα μεταφορών ταυτίστηκαν ως πολύ σημαντικά για την Ένωση στις διαπραγματεύσεις αυτές. Μερικοί από τους ομιλητές δικαίως ανέφεραν ότι μερικά από τα θέματα των μεταφορών θεωρούνται πολύ ευαίσθητα στη ΣΥΠΑ διότι θεωρούνται θέματα εθνικής ασφαλείας, Jones Act κτλ. Ή είναι υπολείμματα νομοθεσίας από το 20 οπότε μπορεί και να ίσχυαν οι περιορισμοί για τις αεροπορικές μεταφορές, για την ιδιοκτησία των εταιριών κλπ. Μπορεί να είχαν και αυτές πτυχές ή βάσεις της εθνικής ασφαλείας, το κατά πόσο αυτό ισχύει ακόμα ιδίως σε διμερείς διαπραγματεύσεις αμφισβητείται. Άρα αντιμετωπίζουμε πράγματι λεπτά πολιτικός θέματα Μερικοί μίλησαν για την τροπολογία Μακέιν που προσπαθεί να καταργήσει το νομοθέτημα Jones Άλλοι λένε ότι θα, θα αποτύχει το εγχείρημα γιατί είχε προσπαθηθεί και στο παρελθόν και δεν πέτυχε. Είναι μια περιοριστική και προστατευτική διάταξη βέβαια που ισχύει και για τις θαλάσσιες και για τις αεροπορικές μεταφορές. Νομίζω λοιπόν ότι καλό θα ήταν να ξαναδείτε τα έγγραφα που έχουμε υποβάλει στο Reading Room αλλά και στις συνόψεις που σας δίνουμε μετά από τους πρώτους αυτούς μήνες των πρωτεύσεων θα έχετε καταλάβει ότι αφιερώσαμε πολύ χρόνο και πολιτικό κεφάλαιο. Δεν έχουμε όμως ακόμη καταλήξει σε καμία συμφωνία ή συνένεση με τη ΣΥΠΑ ως προς την άρση των περιορισμών. Γι' αυτό πιστεύω ότι θα χαρακτήριζα αυτά που είπε ο πρόεδρος έτσι. Υπάρχουν ακόμη και παραδοσιακοί εμπορικοί φραγμοί. Εδώ στις μεταφορές υπάρχουν κλασικοί φραγμοί. Περιορισμοί στις επενδύσεις, ε, κανόνες για την ιδιοκτησία των εταιριών. κλασικοί κλασικοί φραγμοί. Όχι από τα καινούργια θέματα δεύτερης και τρίτης γενιάς. Jones και το νομοθέτημα Τζόνς είναι κλασικός εμπορικός φραγμός. Δεν επιτρέπεται να κάνετε ορισμένες επιχειρήσεις μεταξύ δύο Αμερικανικών λιμανιών εάν δεν είστε Αμερικανός. Και οι κυβερνητικές προμήθειες επίσης είναι παραδοσιακός φραγμός. Κλείνουν την αγορά και λένε τάδε ποσοστό πρέπει να είναι αμερικανικής ιδιοκτησίας η προέλευση. Κλασικός πολλουστατευτιστικός φραγμός. Επομένως, το να λέμε ότι δεν υπάρχουν φραγμοί παραδοσιακοί, ούτε αυτό είναι σωστό. Συνοψίζω, Εκτιμούμε ιδιαίτερο στο γεγονός ότι η Επιτροπή σας τονίζει τη σημασία των κομμάτων μεταφορών στο TTIP και είμαστε διατεθειμένοι να σας πληροφορήσουμε όποτε θέλετε για τις διαπραγματεύσεις και εγώ αλλά και σε υψηλότερο επίπεδο αν θέλετε και για άλλους τομείς ότι οι υπηρεσίες που είναι ο δικός μου. Νομίζω ότι δύσκολα θα περάσουν αυτά που θέλετε στη ΣΥΠΑ. Αλλά και εσείς στις επαφές σας γνωρίζετε, είδατε τι σημασία έχει το θέμα αυτό και πολιτικά. Πολύ δύσκολο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο Βίμ έχει το τελικό λόγο τώρα. Ε. Θέλω να ευχαριστήσω κύριε Πρόεδρε όλους αυτούς οι οποίοι έχουν λάβει το λόγο από τους συναδέλφους μου και την Κομισιόν. Ευχαριστώ. Πρέπει να πάμε το Φεβρουάριο όλες τις Ηνωμένες Πολιτείες για να δούμε με σαφήνεια πώς θα προχωρήσουν τα πράγματα με την συμφωνία TTIP Άκουσα ότι είναι δύσκολο να επανέλθουμε στα γενικά θέματα, όπως είπε και ο κύριος ε, Λάιφριντ όμως. Εγώ νομίζω ότι δεν κάναμε αυτό το οποίο έπρεπε, γιατί τότε ακόμα ήταν τελείως μυστικές οι διαπραγματεύσεις. Εγώ ευτυχώς είμαι μέλος της Επιτροπής ΣΥΝΤΑ και όλα αυτά τα οποία ελέγχθησαν εδώ θα τα μεταφέρω στην Επιτροπή ΙΝΤΑ Χαίρομαι που με <clears throat> συγχαίρουν, αλλά αυτό μου οδηγεί και, με οδηγεί και σε υποψίες. Εγώ είμαι, προτιμώ να είμαι επιφυλακτικός και να μη χαίρομαι πάντα. Για όλα αυτά θα περιμένω τις τροπολογίες που καταδεθούν. Στρέφομαι προς τους συναδέλφους μου, τους φιλελεύθους. Νομίζω ότι είναι απαραίτητο να έρθουμε σε επαφή με την κυρία Μάλστομ ως Επιτροπή Μεταφορών για να τονίσουμε και τον πολιτικό χαρακτήρα, το σημαντικό χαρακτήρα που έχουν οι μεταφορές. Εγώ είμαι λιγάκι παλιωμοδίτικος. Με ενδιαφέρει να μιλήσω με τους ε, διαπραγματεύτες. Πιστεύω ότι από τη μια μεριά πρέπει να υπάρχει κομισιόν, από την άλλη μεριά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μη συγχαίουμε τα δύο. Θα ήταν πολύ χρήσιμο λοιπόν να μιλήσουμε με την κυρία Μάλστον για να αντιμετωπίσουμε τις διάφορες αυτές ερωτήσεις που συζητήσαμε εδώ. Θα ήταν πολύ θετικό. Άκουσα πολλές ε, ε εκφράσεις, διαφάνεια, ανοιχτή εθέρες, πρότυπα, αμοιβαιότητα. Και εγώ χαίρομαι για τις τροπολογίες οι οποίες θα κατατεθούν. Μας λέει η Κομισιόν να πάμε στο δωμάτιο ανάγνωσής της και ίσως πρέπει να πάμε όλοι να το δούμε. Ευχαριστώ λέει και ο αλλά μέχρι στιγμή δεν έχουν μπει όλοι και δεν έχουν δει όλοι τα έγγραφα ακόμα. Μπορούν να πάνε όλοι. Εντάξει. 5 Φεβρουαρίου το μεσημέρι είναι η προθεσμία για τις τροπολογίες. Και κλείνουμε λοιπόν την δημόσια συνεδρία και περνάμε στην συνεδρίαση των συντονιστών και συντονιστριών.